Καλημέρα. Λέω ο Πρόεδρος. Δεν ήταν εύκολο να προσαρμόσουμε την συνεδρίασή μας Τώρα τα καταφέραμε, οπότε τις επόμενες τρεις ώρες θα είμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε την ακρόασή μας. Ακρόαση που έχει να κάνει με την εικαζόμενη παράνομη κράτηση και την μεταφορά κρατουμένων στην Ευρώπη από την CIA. Η ακρόαση αυτή οργανώθηκε στα πλαίσια μιας ε, έκθεσης πρωτοβουλίας ε, μετά από το έργο της Προσωρινής Επιτροπής για την ε, εικαζόμενη παράνομη κράτηση και μεταφορά κρατουμένων στην Ευρώπη. Στόχος είναι να αξιολογήσουμε την κατάσταση, να αξιολογήσουμε τις νέες πληροφορίες που έχουμε και τις εξελίξεις στα κράτη-μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στόχος της ακρόασης αυτής είναι να συνεισφέρει ώστε η δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αναλάβει τις ευθύνες του στα πλαίσια της συνθήκης της, Λισαβίνη, στις Λισαβόνας για τα θεμελιώδη δικαιώματα να γίνει πραγματικότητα. Οι πληροφορίες λοιπόν που έχουμε Οι πληροφορίε λοιπόν που έχουμε όσον αφορά το αίτημα που περιλαμβάνεται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 14 η Φεβρουαρίου του 2007 έχει να κάνει με πληροφορίες που μας έχουν έρθει από μη κυβερνητικέ οργανώσεις, από απλούς πολίτες και όχι από επίσημες πηγές. Γι' αυτό και χαιρόμαστε που σήμερα έχουμε εδώ νομικούς εμπειρογνώμονες και ειδικού ώστε να συζητήσουμε μαζί τους και θα χωρίσουμε τις παρουσιάσεις σε τρία μέρη. Μετά από κάθε τμήμα παρουσιάσεων θα έχουμε συζήτηση. Εννοείται ότι υπάρχει και κάποιο χρονοδιάγραμμα, έτσι, περιορισμένος χρόνος. Γι' αυτό παρακαλώ κάθε ομιλητής να μιλήσει τρία λεπτά περίπου. Μιλάω για τους ευρωβουλευτές που θα έχουν ερωτήσεις, παρατηρήσεις αφού θα έχουμε ακούσει προηγουμένως τις παρουσιάσεις των προσκεκλημένων μας. Σας καλωσορίζω εδώ όλους. Προκαταρτικές παρατηρήσεις όμως θα ακούσουμε από την εισηγήτριά μας για την έκθεση πρωτοβουλίας, την κυρία Ελέν Φλότρο. Θα μας παρουσιάσει το έγγραφο εργασίας το οποίο οδήγησε στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μετά την κυρία Φλότρο θα ακούσουμε τις διάφορες παρουσιάσεις των προσκεκλημένων μας. Παρακαλώ κυρία Φλότρο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Είμαστε εδώ σε αυτή την ακρόαση που έχει να κάνει με την έκθεση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ που αποφάσισε από κοινού με την Υποπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά τα όσα γνωρίζουμε από την έκθεση ΦΑΒΑ. Η έκθεση ΦΑΒΑ, όπως θα γνωρίζετε, είναι μια έκθεση που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2007 μετά από ένα, τε, ένα έτος εργασιών της προσωρινής επιτροπής για το πρόγραμμα το σχετικό της CIA που έγινε με τη συνενοχή χωρών μελών της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και οδήγησε σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, απαγωγές, ε, βασανισμοί, μυστικές κρατήσεις, ανήκουστες παραβιάσεις οι οποίες φυσικά και ε, παραβιάζουν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών αλλά και το διεθνές δίκαιο. Όταν λοιπόν οι, οι εικασίες αυτές ακούστηκαν ήδη από το 2005 και γράφτηκαν στον τύπο σε περιφερειακό ευρωπαϊκό επίπεδο υπήρχαν διάφορες αντιδράσεις. Και εδώ πρέπει να πούμε μπράβο στο ε, Συμβούλιο της Ευρώπης που με τον εισηγητή Martin αλλά και με τον ε, Επίτροπό του για τα ανθρώπινα δικαιώματα πολλές φορές δούλεψαν πάνω σε αυτό το θέμα. Ο Dick Martin εκπώνησε έκθεση, για παράδειγμα, ήδη από το 2005 και έτσι και άρχισε η όλη διαδικασία για να οδηγηθούμε στην έρευνά μας. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, παρενέβη ξανά και ξανά. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το Συμβούλιο, το Ηνωμένο Βασίλειο είχε την Προεδρία τότε, ήρθε σε επαφή με την Κοντολίζα Ράις και βάσει της ικανοποίησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά από τις απαντήσεις της Κοντολίζα Ράις άρχισε το έργο τη η Επιτροπή μας αυτή προσωρινή υπό την Προεδρία του κυρίου Κοέλιου που είναι εδώ και τον ευχαριστώ πολύ για το εξαίρετο έργο τη επιτροπή αυτή. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Φάβα και όλα τα μέλη της προσωρινής αυτής επιτροπής, οι οποίοι δούλεψαν σκληρά. Βλέπω εδώ διάφορα μέλη της προσωρινής αυτής επιτροπής. Καλώς ήρθατε. Στο τελικό ψήφισμα τώρα, στο τελικό κείμενο της έκθεσης ΦΑΒΑ αναφέρεται το εξή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα κράτη-μέλη, θέλει να γίνουν έρευνες ανεξάρτητες από τα κράτη-μέλη για τις εικαζόμενες αυτές παράνομες κρατήσεις και φυλακίσεις και θέλει να αναλυθούν πρωτοβουλίες, οπότε ζητάει από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να βοηθήσουν, να ακολουθήσουν και να πλαισιώσουν τις πρωτοβουλίες αυτές με την δημιουργία μιας ειδικής επιτροπής και είχαμε βέβαια πολλές δυσκολίες και εμπόδια επειδή βέβαια οι διάφορες έρευνες ήταν πάντα περιορισμένες είτε στα κράτη-μέλη είτε στα θεσμικά όργανα αλλά ακριβώ επειδή ήταν ατελής η έρευνα αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να αναλάβει το ίδιο το έργο αυτό μέσω μιας έκθεσης πρωτοβουλίας. Αντίθετα με αυτό που ακούμε συχνά και θα το δούμε και από στις παρουσιάσεις των εμπειρογνωμόνων μας, από τότε έχουμε μάθει πολλά. Η έκθεση ΦΑΒΑ, για παράδειγμα, δεν αναφερόταν σε ε, κρυφές φυλακές στην Ευρώπη. Τώρα πια είναι κάτι που μερικές φορές μάλιστα και έχει αναγνωριστεί στο υψηλότερο δυνατόν επίπεδο, ύπαρξη δηλαδή τέτοιων μυστικών φυλακών. Συνεπώς, σήμερα πια έχουμε ε, νέες πληροφορίες, γεγονότα, πάνω στα οποία μπορούμε να βασιστούμε για να προχωρήσουμε στο έργο μας. Ένας από τους στόχους εξάλλου του εγγράφου εργασίας που έχετε στη διάθεσή σας είναι να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τι εμπόδια έχουν μπροστά τους τα κράτη-μέλη όταν προσπαθούν να βρουν την αλήθεια. Είναι πολιτικά, λείπει η πολιτική βούληση, ή είναι άλλα εμπόδια τα οποία θα μπορούσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να βοηθήσουμε να ξεπεραστούν. Εντοπίζοντας τα εμπόδια αυτά, θα μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να προχωρήσουν οι έρευνες και να ε, δει ε, το φως η αλήθεια. Θυμάμαι ότι ο Ντίν Μάρτιν στην έκθεσή του έλεγε για το πρόγραμμα της CIA με τη Συνολική των Κρατών Μελών τη Ένωση, έλεγε ότι αν ε, μπει αυτό ως πολιτικό μέτρο στην ιστορία που ε, παραβιάζει απαραβίαστα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να παραμείνει σαν ένα απλό γεγονός για το οποίο ποτέ δεν μάθαμε την αλήθεια και για το οποίο ποτέ δεν προσπαθήσαμε να βρούμε ευθύνες. Έχουμε το δικαίωμα αλλά και το χρέος, το καθήκον να μάθουμε την αλήθεια, να επικρίνουμε τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν στο όνομά μας για να προστατεύσουμε την κοινή μας ασφάλεια. Νομίζω ότι αυτό συνοψίζει πάρα πολύ καλά το τι διακυδεύεται στο έργο που θα μαζί να αναλάβουμε. Θα δώσω τώρα πίσω το λόγο στον Πρόεδρο για να μιλήσουν οι προσκεκλημένοι μας. Το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε τόσο ε, εμπειρογνώμ, τόσους πολλούς ε, σημαντικούς εμπειρογνώμονες εδώ, οι οποίοι συλλέγουν πολύτιμες πληροφορίες για μας. Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν είναι εδώ, θα τα πει αυτά και ο πρόεδρος. Εμείς όμως προσκαλέσαμε τις διάφορες αρχές, είτε κρατικές, είτε δικαστικές, είτε κοινοβουλευτικές, που πρέπει να φέρουν σε πέρας κάποια έρευνα στις διάφορες χώρες. Κάποιοι μας είπαν ότι δεν μπορούν να έρθουν εδώ να μιλήσουν μπροστά στους ευρωβουλευτές και μερικές φορές επιχειρηματολογούν. Θα σας διαβάσει τις επιστολές τους και ο Πρόεδρός μας. Μερικές φορές αναλύουν και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούν να είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Πράγμα για το οποίο λυπούμαστε ιδιαίτερα. Τώρα θα ξεκινήσουμε και πρώτα σας παρακαλώ να μου επιτρέψετε να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε καλέσει ομιλητές να συμμετάσχουν στις παρουσιάσεις αυτές ε, εν ονόματι των κρατών μελών και των ε, ε, ε, και ε, προέρχονται από τον ε, δικαστικό και τον κοινοβουλευτικό χώρο. Αλλά μας είπαν ορισμένοι ότι δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν ή στην ακρόαση, οπότε στο τελευταίο τμήμα θα υπάρξει μία εξέταση των ε, απαντήσεών τους στην πρόσκληση και ε, θα ε, σχολιάσουμε τα τις απαντήσεις τις οποίες έχουν υποβάλει προς εξέταση σε αυτή την Επιτροπή. Καταρχήν λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Τζούλια Χολ η οποία είναι η υπεύθυνη για την αντιτρομοκρατία στην Ευρώπη και της δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ την ε, ε, την Επιτροπή που οργάνωσε αυτή την ακρόαση και με κάλεσε να μιλήσω διότι σήμερα έχουν περάσει πέντε χρόνια από την έκθεση του 2007 ε, για τις ε, κρατήσεις ε, ατόμων σε ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA. Οπότε ε, ε, πρέπει να δούμε ποια ήταν η εμπροκή της Ευρώπης στο θέμα αυτό για να προσπαθήσει να επιτύχει μία δυνατότητα να απολογηθεί ε, και να ε, ε, εξηγήσει. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι δεν, υπήρξαμε υπόλογοι, δεν υπήρξαν υπόλογοι οι Αμερικανοί στο θέμα αυτό από το 2007 και θα πω ορισμένα λόγια για τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών και γιατί αυτή η έλλειψη υπευθυνότητος έχει πλήξει και τα θύματα και έχει ε, επηρεάσει και πολλές κυβερνήσεις ε, να προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως αυτές οι οποίες συμμετείχαν στην Αραβική Άνοιξη. Πρέπει να πω ότι άπαξ και ε, δεν, ε, ότι δεν υπάρχει κυβερνητική εκπροσώπηση εδώ και στο τέλος ο πρόεδρος θα μας εξηγήσει γιατί απουσιάζουν. Πρέπει λοιπόν καταρχήν να αντιμετωπίσουμε το συνήθες ε, παράπονο ότι δεν έχουμε να πούμε κάτι νέο σχετικά με τις ενέργειες της CIA στην Ευρώπη. Ε, και όμως αυτό δεν είναι σωστό. Πολλά στοιχεία είναι νέα από το 2007 και ακόμη περισσότερα την τελευταία διετία. Και αυτή η πληροφόρηση ε, μας καλύπτει ορισμένα σημεία του παζλ και παρουσιάζει τη γενικότερη εικόνα της Ευρώπης σε αυτά τα προγράμματα. Ε, Γενικώ όμως θα δείτε ότι υπήρξε προθυμία από τα κράτη-μέλη να ε, παρακολουθήσουν τις κινήσεις αυτές και να ε, απολογηθούν. Ε, υπήρχε μία συνεχής παρουσίαση διαφόρων κινήσεων συμμετοχής και συνενοχής κατά την εξέλιξη των επιχειρήσεων. Διότι το 2009 η ε, Λιθουανία ανεγνώρισε ότι είχε δύο κέντρα κρατήσεων ε, και ε, είχε ζητηθεί από την λιθουανική κυβέρνηση να προβεί σε μία πλήρη έρευνα. Η έρευνα ξεκίνησε το 2010 και σταμάτησε από το το 2011 παρόλες τις πιέσεις των διεθνών οργανισμών που ζητούσαν διάφορες πληροφορίες για τις κρατήσεις και για διάφορες άλλα θέματα τα οποία ποτέ δεν απαντήθηκαν. Οπότε ε, υπήρξε ε, μία ε, συμμετοχή του Γενικού Εισαγγελέα του Δημοσίου Κατηγόρου της χώρας και ζητήθηκε από τις αρχές της Λιθουανίας να ξανανοίξουν αυτή την έρευνα, πράγμα το οποίο η κυβέρνηση αρνήθηκε. θεώρησε ότι τα απορίσματα δεν επαρκούν σαν για να προχωρήσει αυτή η έρευνα. Επίσης υπάρχει μία ανάλυση των στοιχείων σε σχέση με τα προγράμματα αυτά κρατήσεων και παραδόσεων στις Αμερικανικές αρχές και πιστεύαμε στην αρχή ότι στοιχεία τα οποία τότε δεν, ήταν, δεν φαινόντουσαν σημαντικά είναι σημαντικά τώρα λόγω των συνδυασμών τους οποίους έχουμε αποκαλύψει. Και αναφέρω περί ένα παράδειγμα. Όταν η Διεθνής Αμνηστία είπε στις Φιλανδικές Αρχές ότι υπήρχε σύνδεση με μεταξύ της φιλανδικής κυβερνήσεως και των λουαθινικών αρχών σχετικά με τις κρατήσεις αυτές. Ε, τα στοιχεία αυτά δεν είχαν αποκαλυφθεί την πρώτη φορά ε, που συγκεντρώθηκαν το 2006 και μέχρι σήμερα η Φιλανδία έχει αρνηθεί να κάνει την ε, λεπτομερή έρευνα που θα επιτρέψει την αποκάλυψη της αλήθειας και ε, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα υπάρξει μία πλήρης ε, ε, αποκάλυψη. Επίσης όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ της Λιθουανίας και της Δανίας που είχαν εμφανιστεί στα στοιχεία της κοινοβουλευτικής έρευνας στη Λιθουανία το 2009 βλέπουμε ότι ε, το ένα αεροπλάνο ο, ε, η διαδρομή ενός αεροπλάνου ήταν συνήθως Βουκουρέστη, Ρουμανία, Παλάγκα, Λιθουανία, Κοπενχάκη, Δανία στις 18 Φεβρουαρίου του 2005 και άρα η Λιθουανία ε, ε, είχε οργανώσει δύο κρυφά κέντρα κρατήσεως της CIA αλλά τα αποτελέσματα της έρευνας στη Δανία που παρουσιάστηκαν το 2011 περιορίζει τις έρευνες ε, στα στοιχεία μέχρι το 2008 και όχι μετά και ε, δεν έχουμε ε, πορίσματα για την περίοδο από το 2007 στο 2012. <coughs> παρόλα αυτά βλέπουμε ότι ένα ε, αεροπλάνο το οποίο φαίνεται να κινεί σε αυτό το πλαίσιο των ε, κρατήσεων και παραδόσεων ταξίδευσε από το Μπέργεν στο Όσλο ε, και χρία αεροδρόμια στη Λιθουανία αλλά οι αρχές της Νορβηγίας θεωρούν ότι η Αμερικανική κυβέρνηση εξασφάλισε ότι δεν υπήρχε τίποτα μεμπτό ε, σε αυτές τις ε, πτήσεις και ε, αυτό η εύκολη αποδοχή των Αμερικανικών διαβεβαιώσεων στις νορβηγικές αρχές απλώς είναι παράλογη. Ε, ε, το θέμα της συνδέσεως της Σκανδιναβίας στις ε, κινήσεις των κρυφών κέντρων κρατήσεως και στις παραδόσεις της CIA έχει μείνει σκοτεινό παρόλο που είναι πολύ σημαντικό. Οι Ρουμανικές αρχές από την άλλη πλευρά επίσης έχουν απορρίψει τη συμμετοχή τους σε αυτές τις επιχειρήσεις της CIA ενώ πρόσφατες πληροφορίες αποδεικνύουν το, το αντίθετο. Το Δεκέμβριο του 2011 τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης είπαν ότι είχαν εντοπίσει ένα κτίριο στο κέντρο του Βουκρεστίου όπου υπήρχε ένα κρυφό κέντρο κρατήσεως που ονομαζόταν λαμπερό φως και αυτή η έκθεση βασίζεται ε, σε διάφορα στοιχεία που διατείνονται ότι η Ρουμανία είχε τουλάχιστον μία κρυφή φυλακή. Ε, είναι βασικό ότι οι πληροφορίες αυτές ε, δεν έχουν ενοχλήσει μέχρι στιγμής ε, τις ουρμανικές αρχές οι οποίες δεν έχουν αντιδράσει και τις θεωρούν ανύπαρκτες και θεωρούν ότι να αρνούνται την ευθύνη τους είναι πάρα πολύ εύκολο παρόλο που κατηγορούνται για συμμετοχή σε αυτές τις επιχειρήσεις της CIA ναι, και από την άλλη μεριά διατείνονται ότι δεν ε, υπάρχει καμία βάση σε αυτούς τους ισχυρισμούς. Στην ε, Πολωνία επίσης ε, υπάρχουν δύο, δύο κρατούμενοι οι οποίοι προσπάθησαν να υπερβούν τα ε, ε, τα στοιχεία και τους περιορισμούς ε, των εθνικών κρατών και να απευθυνθούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ε, βλέπουμε όμως ότι υπήρξε μία ανακοίνωση την οποία δεν έχουμε αναλύσει ακόμη και λέγει ότι θα έπρεπε οι πολωνικές αρχές να έχουν οδηγηθεί σε ε, μία αγωγή, αγωγή στη δίωξη και στην καταδίκη. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχει γίνει τίποτα και τώρα επανέρχομαι στο Ηνωμένο Βασίλειο, διότι τον Ιούλιο του 2010 το Ευρωπαϊκό το, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είχε αναφέρει ότι έγινε μία σημαντική έρευνα αλλά ε, υπήρχε πλήρης ε, κυβερνητικός έλεγχος ε, της αποκαλύψεως των πληροφοριών πράγμα το οποίο οδήγησε τους πρώην κρατουμένους και το, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις να μποϊκοτάρουν τη διαδικασία αυτή και η ε, αποκάλυψη των ε, εγγράφων ε, από το Human Rights Watch στην Τρίπολη απέδειξε ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είχε συνεργαστεί με την CIA και είχε τουλάχιστον παραδώσει τουλάχιστον δύο άτομα και της οικογένειάς του στη Λιβύη το 2004. Ε, υπήρξε λοιπόν μία συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε αυτές τις δραστηριότητες και εις ε, την αντιμετώπιση των κρατουμένων ε, σε ξένες χώρες. Υπάρχουν και πολλά άλλα στοιχεία και το Κοινοβούλιο έχει ψηφίσει το ψήφισμα του 2007 αναφέροντας τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Σουηδία χωρίς όμως να έχει υπάρξει καμία αποκάλυψη στις Ηνωμένε Πολιτείε, διότι ε, το, η κυβέρνηση ο Ομπάμα έχει αποφύγει ε, και απορρίψει όλες τις κατηγορίες. Υπάρχει όμως ε, το, η, η κασική περίπτωση Rich Aviation vs. Spotfire όπου αποδεικνύεται ότι υπήρχαν σχέσεις αναθέσεως και υπεργολαβίας για την παροχή και διάθεση ιδιωτικών αεροπλάνων για την μεταφορά των παρανόμων μετακινήσεων ατόμων από τη CIA διεθνώς και στην Ευρώπη. Υπάρχουν πάρα πολλά τιμολόγια σε αυτήν την δικαστική διαμάχη που αποκαλύπτουν τα στοιχεία και πλέον δεν υπάρχει μυστικό σε αυτό το θέμα. Η ιδέα ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να είναι υπόλογοι όπως άλλωστε και τα άτομα για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, δεν ε, έχει ε, επιτρέψει να ισχύσει η αρχή της, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βλέπουμε παραδείγματο χάρη ότι ο υπουργό Εξωτερικός της Δανίας είχε είχε συντάξει ένα σχετικό άρθρο στην εφημερίδα European Voice της 19 Μαρτίου του 2012 και ε, η αποτελεσματική ε, ε, όπως λέγει αντιμετώπιση των αντιτρομοκρατικών μέτρων και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι αντιφατική στόχη αλλά πρέπει να είναι συμπληρωματική και να ενισχύουν αλλήλεις. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εις τα πλαίσια της ε, ακροάσεως της Επιτροπής σας θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα σταματήσει η ατιμορρησία και δεν θα συνεχιστεί. Ε, το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά κράτη ε, λέγεται ότι έχουν συμπράξει σε τέτοιες απεχθείς, σε τέτοιες παραβιάσεις και παράνομες μεταφορές ε, είναι ατυχές και αυτό διακηρύσσεται στο ίδιο άρθρο της εφημερίδας European Voice. Άρα οι συντάκτες του άρθρου αντιλαμβάνονται ε, και συμφωνούν ότι υπάρχουν, ε, υπάρχει αλήθεια σε αυτές ε, τις αιτιάσεις για παράνομες κρατήσεις και ε, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να στηρίζει και να προωθεί ε, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή στην ε, διεθνή κοινότητα και να συμβάλλει ώστε τα κράτη-μέλη να σταματήσουν τις κινήσεις αυτές και να απολογηθούν πρέπει κατά αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουν και τις ε, νέες κυβερνήσεις των αραβικών χωρών να αναμορφώσουν τον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου στην περιοχή τους. Πώς θα γίνει όμως αυτό αν ε, τα χέρια της Ευρώπης δεν είναι καθαρά και υπάρχουν ε, αιτιάσεις και δικαιολογίες ε, όταν αναφέρεται ότι υπάρχουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εν ονόματι της αντιτρομοκρατίας. Ζητούμε λοιπόν να υπάρξει μία πλήρη συνεργασία, ε, αποκάλυψη όλων των πληροφοριών, να επισκεφθούμε ε, τους χώρους κράτησης και όπως είχε συμφωνηθεί στο ψήφισμα του 2007 να υπάρχει μία αμερόληπτη έρευνα στις ε, αιτιάσεις συμμετοχής της Ευρώπης στα προγράμματα αυτά κατά τρόπον ώστε να μπορέσει να, δοθεί, ε, να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα αυτών των κινήσεων και να εξασφαλίσουμε ότι ε, οι εξάρσεις, οι βασανισμοί που συνεπάγονταν αυτές οι παράνομες κρατήσεις δεν θα ξανασυμβούν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κυρία Χολ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Θα θέλαμε να, ακούσουμε τώρα τη δεύτερη παρουσίαση του κύριου Κρόφτον Μπλακ, που είναι ερευνητής για τις μυστικές φυλακές και τις απαγωγές κρατουμένων και τις μυστικές πτήσεις, μέλος της, της Reprieve. Κύριε Μπλακ, έχετε το λόγο και μετά θα δώσουμε το λόγο στα μέλη που θα σας θέσουν ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Τζούλια, για την πολύ ε, εφραδή παρουσίασή σου. Θα ήθελα να σας δώσω λίγα στοιχεία για τις νέες πληροφορίες που προέκυψαν μετά από έρευνες της Reprieve και από άλλες ε, οργανώσεις. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τα δεδομένα των πτήσεων, καταρχάς. Από το 2007 ε, έχουμε όλο και περισσότερες πληροφορίες για τις α, πτήσεις αυτές και το δίκτυο των πτήσεων. Έχουμε βρει νέα αεροπλάνα. Μπορέσαμε να επαναξιολογήσουμε τη σημασία των αεροπλάνων που είχαμε βρει, για το οποία είχαμε βρει στοιχεία πριν και πολλές, ε, πολλοί από τους μετέχοντες από την ε, συνεδρίαση παίξαν σημαντικό ρόλο από τη Διεθνή Αμνηστία, από τη Reprieve, από την Access Info Europe. Ε, πολλοί έχουν κάνει τις δικές τους έρευνες, ορισμένοι πιο, με περισσότερο ζήλο από άλλους για την δουλειά που έκανε η Republic Access Info Europe. Θέλω να σας πω ότι ε, κάποιες κυβερνήσεις έχουν κάνει κάποια προσπάθεια, όπως η Δανία, η Φιλανδία, η Λιθουανία και άλλες, για να δώσουν στοιχεία και να βρουν πληροφορίες. Ε, δεν είναι παρκής όμως αυτές, γιατί είναι κατακαιρματισμένες. Ε, δεν αρκεί να βρούμε ε, κάποια στοιχεία για το που πέρασε η πτήση. Δεν μας δείχνει ακριβώς την, την ολότητα του δικτύου. Ε, γιατί τα αεροπλάνα αυτά, τα μυστικά αυτά αεροπλάνα κάναν πάρα πολλέ στάσεις για να, ανεφοδιασμό, για να στά, ε, σπάσουν το ταξίδι, ε, για να μην αποκαλυφθεί το ταξίδι. Και με πολύ αργό τρόπο βρίσκουμε στοιχεία, βρίσκουμε ψηφίδες του παζλ για τις χώρες από τις οποίες πέρασε το αεροπλάνο. και όλα αυτά τα στοιχεία τα έχει στη διάθεσή της μία εταιρεία, το Eurocontrol. Η Ριπρίβ προσπάθησε με τη βοήθεια άλλων να βάλει όλα μαζί τα στοιχεία αυτά Υπάρχουν πάρα πολλά κενά ακόμα, παρότι έχουμε αρκετά στοιχεία πια, ε, και αυτό οφείλεται στην προθυμία πολλών ευρωπαϊκών χωρών να απαντήσουν στα αιτήματα για πρόσβαση σε πληροφορίες. Από την έκθεση που ε, που γράψαμε ε, πέρυσι ε, προκύπτει ότι από τις 28 χώρες ε, με τις οποίες ήρθαμε σε επαφές, οι 14 αρνήθηκαν να απαντήσουν. Επομένως, έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε ακόμα. Αυτή τη στιγμή εστιάζουμε στην συνενοχή των εταιριών σε αυτές τις πτήσεις. Υπάρχουν κάποιες νόμιμες εταιρείες που συνεργάζονται με την Αμερικανική κυβέρνηση. Όπως είπε και η Τζούλια, βασικό στοιχείο ήταν η η μήνυση που έγινε στην Αμερική ενάντια στις υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας και όπου έδειξε τη συνενοχή πάρα πολλών αμερικανικών εταιριών ε, με το πρόγραμμα αυτό ε, μυστικών παγωγών, πτήσεων κτλ. Ε, υπάρχουν τράπεζες, υπάρχουν συνταξιδοτικά ταμεία, που εμπλέκονται σε όλη αυτή την επιμελητιακή προσπάθεια του προγράμματος. Το να βρεθούν αεροπλάνα, ε, πληρώματα, να μπουν τα πληρώματα μέσα στα αεροπλάνα, να βρουν το δρόμο, τη διαδρομή, τον ανεφοδιασμό, ε, επικοινωνίες, ε, να στείλουν τα σχέδια της πίσης, να βρουν το χώρο στέγασης για τα πληρώματα των αεροπλάνων αυτών. Ε, σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτές οι πτήσεις έγιναν για ένα πελάτη, την Αμερικανική κυβέρνηση. Από τις τηλεφωνικές πληροφορίες αποκαλύπτεται ε, ένα μοντέλο συμπεριφοράς γύρω από αυτές τις πτήσεις, ένα μόντους απεράντη. Από, τα, από την τεράστια τεκμηρίωση που έχουμε φαίνεται ε, πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο τελικός ανάδοχος είναι η Αμερικανική κυβέρνηση. Οι εταιρείε αυτές γενικά που οργάνωσαν αυτή την ε, προσπάθεια δεν είναι ευρωπαϊκές εταιρείε, αλλά ε, πούμε η δανέζικη κυβέρνηση ε, έλαβε χρήματα από αεροπλάνα τα οποία πέρασαν από πάνω ε, με σκοπό τη μεταφορά σε μυστικές φυλακές. Η δουλειά που κάνει η η Reprieve είναι να συνδέσει όλες αυτές τις συναλλαγές με τις μεταφορές κρατουμένων. Μερικές φορές δεν είμαστε ε, σίγουροι. Ε, ορισμένα αεροπλάνα ε, δεν μετέφεραν τους φυλακισμένους, αλλά άλλους που εμπλέκονται στο δίκτυο, ας πούμε, με μεταφραστές ανακριτές κτλ. Ε, όλες, όλες αυτές οι πτήσεις είναι ζωτικό στοιχείο του δικτύου. Ε, από την τελευταία φορά που σας ε, επισκέφτηκα ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βρήκαμε δύο μυστικές φυλακές στη Λιθουανία και στη Ρουμανία. Τα βρήκαν αυτά τα στοιχεία δημοσιογράφοι και αυτές οι αποκαλύψεις και στις δύο περιπτώσεις συνοδεύονται από άφθονη τεκμηρίωση. Η φυλακή στη Λιθουανία είναι σε ένα χωριό κοντά στο Βίλνιους. Μία μυστή εταιρεία ε, αγόρασε αυτό το μέρος και το έδωσε σε ένα άτομο. Το 2000, τον Ιούλιο του 2003 και τον Μάρτιο του 2004 ε, το άτομο αυτό αγόρασε από ντόπιου ε, το χώρο και μίλησε για ένα πρόγραμμα κατασκευής ε, το οποίο ε, το επόπτευαν οι Αμερικάνοι. Ε, πολλά αυτοκίνητα με μαύρα παράθυρα επισκέφτηκαν το χώρο αυτό και τον Ιανουάριο του 2007 πωλήθηκε στους, στις σημερινούς ιδιοκτήτες που είναι οι μυστικές υπηρεσίες της Λιθουανίας. Έχουμε στοιχεία για διάφορες πτήσεις που, και αεροπλάνα που συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα μυστικών πτήσεων που έκαναν έφτασαν στην ε, Λιθουανία, μερικές φορές ε, περνώντας από την ε, Φιλανδία και τη Σουηδία για να μην αποκαλύψουν τη διαδρομή. μία άλλη πήγε από τη Λιθουανία στην Πορτογαλία και μετά στην Αίγυπτο. Επίσης, οι μυστικές υπηρεσίες έδωσαν εντολές στους συνοριοφύλακες να μην διενεργήσουν τους κλασικούς ελέγχους. Ε, τίποτα δεν έγινε με το φυσιολογικό τρόπο. Ε, αυτά τα αεροπλάνα επίσης επισκέφτηκαν τη Ρουμανία. Ε, έχουν γίνει και άλλες, έγιναν και άλλες τάσεις από διάφορα αεροπλάνα. Και έχουμε στοιχεία ότι όλες αυτές οι πτήσεις συνδέονται με την ε, ανάδοχο εταιρεία και τελικά με την Αμερικανική κυβέρνηση. Ξέρουμε ότι ε, η CIA ε, στα βορειοδυτικά του Βουκουρεστίου είχε μία φυλακή κάτω από το Γραφείο Κρατικών Αρχείων για απόρτες πληροφορίες. Εκεί κρατούνταν διάφοροι φυλακισμένοι. Ε, έγιναν κάποιες έρευνες για αυτό το θέμα και έχουμε πολύτιμα στοιχεία. Όμως, δυστυχώς, ε, η ποιότητα αυτών των στοιχείων ε, δεν αξιοποιείται γιατί δεν βγαίνουν τα σωστά συμπεράσματα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει άλλες ερμηνείες, χρησιμοποιεί διάφορες, διάφορα σημειολογικά στοιχεία και τα πορίσματα της έρευνας του 2009 ε, λένε ότι λένε μάλλον οι Ρουμάν, οι αξιωματούχοι, ότι αυτό είναι θέμα ερμηνεία. Εγώ, είπε κάποιο ε, Ρουμάνο αξιωματούχο, δεν κράτησα κανέναν τρομοκράτη από το χεράκι, επομένω δεν μπορώ να σα δώσω απαντήσει. Ε, τέτοιου είδου απαντήσει τι δίνουν όλε αυτέ οι χώρε που εμπλέκονται. Και αν κάποιες, κάποια στοιχεία υπάρχουν, προσπαθούν να βρουν τρόπους διαφυγής. Ας υποθέσουμε ότι δεν υπήρξαν τέτοια προγράμματα, δεν υπήρξαν μυστικές φυλακές. Α, ας ενώσουμε τις τελίτσες αυτές και τις ψηφίδες του παζλ για να δούμε πώς συνέβη κάτι άλλο. Όμως η... αυτό που προκύπτει είναι ότι είναι μάλλον απίθανο. Ένα παράδειγμα. Στην προδικαστική έρευνα οι Λιθουανοί ε, ανακριτές βρήκαν ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που μας δείχνει ότι κάποιος κρατήθηκε μυστικά στη Λιθουανία. Ε, όμως δεν έχουν τη δυνατότητα να εξηγήσουν πώς υπάρχουν όλα αυτά τα ε, κτίρια στη Λιθουανία. Δεν είναι κατά ανάγκη φυλακές μας είπαν. μπορεί να δημιουργήθηκαν για να βάλουμε τη μαλφή τι είναι αυτά τα τιμαλφή τα οποία ε, έπρεπε να κρύψει σε ένα μικρό χωριό η Αμερικανική κυβέρνηση έξω από το Βίλνιου. Ε, να φτιάξει ένα κτίριο, ειδικά κατασκευασμένο που το επόπτευαν οι Αμερικανικές ε, ε υπηρεσίες και που πηγαινοέρχονταν έρχονταν αυτοκίνητα με μαύρα παράθυρα. Ε, για ποιο λόγο πήγαν Αμερικανοί στο Βουκουρέστι, στη Ρουμανία, τι είδους τιμαλφή έκρυβαν εκεί. Διάφορες χώρες έκαναν έρευνες για το ρόλο τους ε, σε αυτά τα προγράμματα και για να συγχωρεθούν ε, είπαν ότι δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξει ότι υπήρχαν ε, φυλακές για αυτά τα αεροπλάνα. Αυτό είναι αβάσιμο. ήταν, πρόκειται για μια παγκόσμια συνωμοσία της Αμερικανικής κυβέρνησης. υπήρχε ένα τεράστιο δίκτυο με τη συνοχή εταιριών, κυβερνήσεων κτλ έπρεπε διάφορα άτομα να τα πετάξουν, όχι μόνο τους φυλακισμένους, αλλά ανακριτές, ε, ε, μεταφραστές κτλ. Όλα αυτά τα άτομα ήταν σημαντικά για το δίκτυο. Διάφορες χώρες, το Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία, Ισλανδία, ε, έπαιξαν ένα στρατηγικό ρόλο σε αυτό το δίκτυο. Ε, χωρίς να υπάρχουν στις επικρατείες τους μυστικές φυλακές. Άλλες χώρες επισκέφθηκαν πιο σπάνια στα πλαίσια αυτού του προγράμματος. Καταλήγοντας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή είναι σε στεναρή θέση. Μπορεί να αξιοποιήσει την πρόοδο που έγινε. Αλλά για να υπάρξει πρόοδος πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι μυστικές φυλακές και αυτά τα προγράμματα πτήσεων, απαγωγών και πτήσεων υπήρξαν. Και πρέπει να δούμε ακριβώς ποιο συμμετείχε σε αυτό το δίκτυο. Θα πρέπει επίσης να ελέγξουμε τη συμπεριφορά διαφόρων κυβερνήσεων και να δούμε κατά πόσον είναι βάσιμες οι οι αρνήσεις τους. Ε, είναι πιθανά αυτά που λένε, ε, λαμβάνουν υπόψη τα στοιχεία. Ε, στη Ρουμανία και στην ε, Λιθουανία, παρά τις αρνήσεις, αποδείχτηκαν ότι λέγαν ψέματα. όλα αυτά τα στοιχεία δεν προέκυψαν από τους εισαγγελείς, αλλά από τους α, ανεξάρτητους ερευνητές. ψηφίδα-ψηφίδα, βήμα-βήμα και είναι αντιπαραγωγικό να μιλάμε για ισχυρισμούς ε, για αυτό το θέμα. Εκτός και αν μιλάμε για πολύ συγκεκριμένα στοιχεία όπου πραγματικά υπάρχουν αβεβαιότητες. Ε, αλλά κατά τα άλλα έχουμε στοιχεία, έχουμε αποδείξεις, έχουμε τεκμήρια. Δεν πρόκειται για ισχυρισμού. Αύριο, 28 Μαρτίου, είναι η επέτειος της ε, σύλληψης του Αμπού Ζουμπαϊντά, που ένα άτομο το οποίο ε, ήταν σημαντικό για το πρόγραμμα αυτό και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη της, του όλου δικτύου. Ε, ελπίζω να μην να ε, τους ξεχάσουμε. Thank you, Mr. Black. Now... Ευχαριστούμε κύριε Μπλακ. Συζήτηση τώρα. Σας υπενθυμίζω ότι προκειμένου να καταφέρουμε με τον χρόνο που έχουμε να ακούσουμε όλους τους προσκεκλημένους μας, έτσι καλλιώς στις 12 πρέπει να έχουμε τελειώσει με την ακρόαση αυτή, καλό θα ήταν οι ερωτήσεις σας να περιορίζονται παρακαλώ σε τρία λεπτά που έχει ο καθένας σας. Έτσι οι προσκεκλημένοι μας θα μπορέσουν και να απαντήσουν σε ό,τι ερωτήσεις έχετε. Αρχίζουμε με την κυρία Άννα Γκόμες. Αλλά δεν είναι εδώ. Η κυρία Ινχετφέλτ τότε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση. Το συζητάμε τόσα χρόνια αυτό το θέμα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αντιλαμβάνομαι φυσικά την απογοήτευση και των δύο ομιλητών, κυρίως της κυρίας Χολ. Αναρωτιόμαστε τι θα μπορούσε να γίνει παραπάνω γιατί δεν νομίζω ότι εμείς έχουμε ούτε τη δυνατότητα, αλλά ούτε και την εντολή να κάνουμε εμείς τις έρευνες. Είναι δουλειά της αστυνομίας να κάνει ανακρίσεις, δεν είναι δικιά μας δουλειά. Και έπειτα υπάρχουν τόσα πολλά γεγονότα, είναι σαν ένα γίγα παζλ με χίλια κομμάτια και λείπουν τα δέκα. Την εικόνα τη βλέπουμε παρόλα αυτά. Οι χώρες μέλη δεν φαίνεται να αρνούνται πια τα γεγονότα αλλά δεν λογοδοτούν βέβαια, σιωπούν. Ο Τιν Μάρτιν νομίζω το αναφέρει κάπου ότι πρόκειται για τον τοίχο της σιωπής. Είναι ντροπή. Και γιατί τα καταφέρουν έτσι, γιατί σιωπή η κοινή γνώμη τελικά. Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να βρεθούν αντιμέτωποι με μια δικιά του εικόνα, η οποία να είναι τελικά κάπως διαφορετική από εκείνη που πίστευαν ότι ήταν η πραγματική όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς αποφεύγουμε λοιπόν να μάθουμε ότι είμαστε συνυπεύθυνοι για τα γεγονότα αυτά. Έχω όμως να ρωτήσω και κάτι. Επικεντρωνόμαστε πάντα σε συγκεκριμένες χώρες. Λέμε Πολωνία, Λιθουανία, Ρουμανία. Εντάξει, είναι και αυτό το πρόβλημα, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει συλλογική ευθύνη επίσης. Υπάρχει συλλογική ευθύνη γιατί τότε οι υπουργοί το συζήτησαν και μπορεί να μην είναι υπεύθυνοι. Εντάξει, στη χώρα μου δεν νομίζω ότι υπάρχουν ε, μυστικές φυλακές, αλλά η χώρα μου σίγουρα το ήξερε το πρόγραμμα, οπότε είναι συνυπεύθυνοι. Και νομίζω ότι όλες οι χώρες είναι συνυπεύθυνε. και θα έπρεπε να τις αφορά η έκθεση αυτή όλες. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι ζούμε στην εποχή του διαδικτύου. Έχουμε το Wikileaks. Αν ναι, οι χώρες ε, δεν θέλουν το Wikileaks, ας φροντίσουν οι ίδιες να προσφέρουν περισσότερη διαφάνεια. Ας τα εξηγούν οι ίδιες οι χώρες τους πολίτες τους και ας μην περιμένουν ε, το επόμενο που θα βγάλει το Wikileaks. Και εξάλλου, αν επιμένουν για το ότι οι ισχυρισμοί δεν είναι παρά ισχυρισμοί, τότε γιατί φοβούνται την έρευνα. Γιατί αν είναι τόσο σίγουροι ότι τίποτα δεν συνέβη, ε, τότε θα έπρεπε να τη θέλουν την έρευνα γιατί θα τους δώσει την ευκαιρία να αποδείξουν ότι πρόκειται απλώς για ισχυρισμού και τίποτα δεν είναι αλήθεια. Και δύο τελευταία θέματα για την ηθική πτυχή. Δεν μπορούμε να επιμείνουμε ποτέ αρκετά σε αυτό γιατί κάθε μέρα οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν από τον Ασάντ να φύγει από την εξουσία. Το ίδιο κάναμε τον Μουμπάρακ, με τον Καντάφη. Και εμείς επίσης. Ναι, αλλά πριν από λίγα χρόνια εμείς στέλναμε ανθρώπους ακριβώς σε αυτές τις χώρες. Στέλναμε τους ανθρώπους για ειδικέ ανακρίσεις όπως τις λέγαμε, για βασανισμούς δηλαδή. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να ξεχνάμε το δικό μας τον ρόλο σε όλη αυτή την υπόθεση και να λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να εγκαταλείψουν την εξουσία που θα έπρεπε και θα έπρεπε να δικαστούν, δεν λέω. Οπότε και ο κύριος Κερκόβε και άλλοι. Αυτό είναι αρμόδιο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Εκείνος θα μπορούσε να πιέσει για να αλλάξει η κατάσταση. Αν είναι σοβαρός και θέλει όντως να αντιμετωπίσει ε, αυτά τα γεγονότα, μα κύριε Κέρκοφ, εσείς θα έπρεπε να αναλάβετε δράση. Γιατί δεν το κάνετε, γιατί δεν πιέζετε εσεί τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε πραγματικέ έρευνες, αν εννοείτε αυτά που λέτε, εσείς πρέπει να το κάνετε κύριε Κέρκχοφε αυτό. Ευχαριστώ. Ας ακούσουμε πρώτα και άλλες ερωτήσεις και μετά. Η κυρία Μόρμπα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστώ που οργανώσατε αυτή την ακρόαση. Ίσως κάποια στιγμή ξυπνήσω και καταλάβω ότι πρόκειται για ένα κακό όνειρο. Τι γίνεται, είμαστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε εδώ διάφορους εμπειρογνώμονες, με κυβερνητικές οργανώσεις που μιλούν για την κυβέρνηση των Πολιτειών και λένε ότι έχουν ε, ε, διαπράξει σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ε, δικαίου και εγκλήματα, βασανισμούς κλπ. Σε ευρωπαϊκό έδαφος, στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τρεις ερωτήσεις έχω. Πρώτον, είμαι μέλος στην αντιπροσωπεία για τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε το σώμα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε δημιουργήσει αντιπροσωπείες για διακοινοβουλευτικές ε, σχέσεις. Είναι δηλαδή ευρωβουλευτές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίοι επισκέπτονται συχνά τις Ηνωμένε Πολιτείε, το Κογκρέσο εκεί. Και Εκεί συζητούμε διάφορα θέμα. Εγώ είμαι λοιπόν μέλος της αντιπροσωπείας αυτής και εγώ δεν ξέρω να το έχουμε θίξει αυτό διμερός αυτό το θέμα. Τουλάχιστον τελευταία φορά που πήγαμε στις Ηνωμένε Πολιτείε, το ξέρω σίγουρα ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο. Συνεπώς, σε τι χρησιμεύουν οι αντιπροσωπείες ε, αυτές, δεν θα μπορούσαν και αυτές να κάνουν κάτι. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη ναι θα μπορούσαμε να είχαμε ένα κατάλογο με γεγονότα, το τι ακριβώς δηλαδή έχει γίνει μέχρι τώρα. Δηλαδή ποιες είναι οι κυβερνήσεις οι οποίες συμμετέχουν, τι έρευνες έχουν ήδη γίνει από τις κυβερνήσεις αυτές, αν υπήρξαν ε, δεν για τη Ρουμανία, τη Δανία και τα αν υπάρχουν ε, στοιχεία για το τι ακριβώς έχει γίνει γεγονότα δηλαδή, για να ξεχωρίσουμε τα γεγονότα από τις εικασίες. Και το τρίτο, για να απαντήσω στην κυρία Χετβέλτ. Νομίζω ότι εμείς ατομικά, επειδή είμαστε εκλεγμένοι πολιτικοί, και εμείς είμαστε υπεύθυνοι για να ενημερώνουμε τους ε, πολίτες μας, τις χώρες μας. Στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, στη χώρα μου, είμαι σίγουρη ότι ελάχιστοι γνωρίζουν αυτή την υπόθεση, ότι υπάρχουν τόσο σοβαροί ισχυρισμοί για τόσο σοβαρά εγκλήματα. Είναι απίστευτο ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε εξακολουθούν να παίζουν το ρόλο του θεματοφύλακα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να επικρίνουν τη χώρα μου, για παράδειγμα, για πράγματα που έχουν να κάνουν με την προστασία των δεδομένων, με το διαμεσολαβητή, με τα δικαιώματά του κλπ. Δεν είναι περίεργο αυτό κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, η κυρία Γκόμες τώρα που ήρθε. Η σειρά σας κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που οργανώσατε την ακρόαση αυτή και για τις παρουσιάσεις των ε, εμπειρογνωμόνων μας. Σίγουρα είναι αποφασιστική σημασία για το έργο μας. Τώρα άκουσα από την κυρία Μορβάη μην νομίζει, το έχουμε θίξει. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν το έχουμε θίξει στις αντιπροσωπείες στο θέμα αυτό των ε, παράνομων εκδόσεων ε, της CIA. Έχει τεθεί ε, σε συνάντηση με τους αδέρφους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ακριβώς αυτό άνοιξε και το δρόμο για τη δουλειά που έγινε από την Αμερικανική πλευρά που ξεκίνησε επί Μπούς και συνεχίστηκε με τον Ομπάμα, ώστε κάποιοι που κρίθηκαν αθώοι τελικά να ε, μπορούν να φύγουν και να πάνε σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Εγώ ήμουνα στην Επιτροπή αυτή με το ΦΑΒΑ και είναι ζωτική σημασία ε, η δουλειά που έγινε εκεί και που πρέπει να συνεχιστεί υπό το φως των νέων πληροφοριών. Όσον αφορά τη χώρα μου την Πορτογαλία, θυμάμαι ότι στο τέλος των εργασιών της Επιτροπής ΦΑΒΑ πήγαμε στην Πορτογαλία. Εγώ μάλιστα πέρασα ολόκληρη μέρα να ζητάω κατάλογο με πτήσεις από πώς Γουαντάναμο που πέρασαν πάνω από τον ανέριο χώρο της Πορτογαλίας. Μου τα αρνήθηκαν, μου είπαν ότι δεν υπήρχαν. Και όμως κάποια στιγμή έμαθα ότι υπήρχαν. Και μπόρεσα να το συμπεριλάβω στην έκθεση ΦΑΒΑ. Βέβαια δεν το αναλύσαμε ποτέ. Είναι όμως ένα σημαντικό στοιχείο, γιατί αποδεικνύει αυτά που λένε και οι ομιλητές μας εδώ, ότι έγιναν πολλά και ότι υπήρχε σαφέστατα συνενοχή από τις αρχές, οι οποίες στο κάτω-κάτω ή που ήταν εντελώς ανίκανες και τελικά τους ξεγέλασαν, τους κορόιδεψαν οι Αμερικανοί ή ήταν πλήρως συνένοχοι. Και από τη δικιά μου την έρευνα έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για το δεύτερο. Θα ήθελα μια κοινοβουλευτική έρευνα στην Πορτογαλία, όμως ε, δεν έγινε πραγματικότητα, δεν τα καταφέραμε ούτε καν το δικό μου το κόμμα. Και η δικαστική έρευνα που ζητούν που ζητούμε και εμείς, το ζητήσαμε στον Ισαγγελέα, τι έγινε, δύο χρόνια κράτησε, ανακαλύφθηκαν διάφορα πράγματα και ξαφνικά σταμάτησε, έκλεισε. Αγνοήθηκαν όλα τα σημαντικά πράγματα τα οποία αποκαλύφθηκαν και που ήταν πολλά. Και αρκεί κανείς να κοιτάξει τους 13 τόμους που συγκεντρώσαμε σε τρεις μέρες. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για πολλά, για πάρα πολλά, που επίσης μας έχουν ξεφύγει. Έκλεισε η έρευνα αυτή για πολιτικούς λόγους, για κανέναν άλλον για πολιτικούς λόγους, για να μην αποκαλυφθούν άλλα. Οι έρευνες πάντως δείχνουν ότι η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια στα αεροδρόμια της Πορτογαλίας και όχι μόνο και σε άλλες χώρες, η κατάσταση ασφάλειας λοιπόν δεν είναι καλή. Γιατί αν γίνονται τέτοια πράγματα με αεροπλάνα όπως αυτά που λέμε πολιτικής αεροπορίας ε, και μας ξέφυγαν, ε, φανταστείτε τι μπορεί να γίνει και με οποιοδήποτε άλλο αεροπλάνο. Έπειτα, τα αεροπλάνα αυτά φαίνεται ότι περνάνε τη μια μέρα με ένα συγκεκριμένο χρώμα και μια συγκεκριμένη... Ε, με κάτι συγκεκριμένο αναγράφεται σε αυτά, την άλλη μέρα έχουν αλλάξει χρώμα. Ξαναπερνάνε με άλλο χρώμα και με άλλη επιγραφή. Φαίνεται ότι τα αεροπλάνα αυτά της πολιτικής αεροπορίας ζητούν πάρα πολύ πάγο, για παράδειγμα, από τις αρχές. Και αυτό είναι που βρήκανε περίεργο και οι δημοσιογράφοι στα Κανάρια. Γιατί αυτά τα αεροπλάνα πολιτικές αεροπορίες να ζητούν τόσο πολύ πάγο. Τι σημαίνει αυτό, ότι κάποιοι είναι πληγωμένοι ή τι κάτι άλλο μεταφέρανε. Στην περίπτωση της Πορτογαλίας πάντως υπάρχουν δηλώσεις από στρατιωτικούς αξιωματούχους που λένε ότι όλη η διαδικασία ε, άδεια που παίρνουν τα αεροπλάνα αυτά ε, ήταν ε, γνωστή. Ήταν γνωστό δηλαδή ότι υπήρξε ευαίσθητο φορτίο φυλακισμένων. Πάντως επιπλέον από όλα αυτά γιατί δεν πρόκειται μόνο γι' αυτό και δεν ήταν μόνο τα αεροπλάνα της πολιτικής αεροπορίας, αλλά ήταν και στρατιωτικά αεροπλάνα. Και όχι μόνο αμερικανικά, από τη Σαουδική Αραβία υπάρχει στους καταλόγους και βρετανικά και γαλλικά και βελγικά και ελληνικά. Και πρόκειται και για πλοία. Και εγώ το είπα, έδωσα το όνομα του ατόμου στην Πορτογαλία που παρουσίασε μια γνωμοδότηση για την αλλαγή στην αυσιπλοεία για να μην ενοχληθούν τα πλοία αυτά. Τα έχω όλα τα στοιχεία και τα έδωσα το όνομα, τα στοιχεία όλα. Δεν ε, διαψεύστηκαν ποτέ, αλλά δεν συμπεριλήφθηκαν και σε καμία έρευνα. Ειλικρινά, λοιπόν, πιστεύω. Α, ναι και για τι αζόρε τη Πορτογαλίας και την βάση εκεί. Υπάρχουν μαρτυρίες που τις έχω που είπαν ότι είδαν φυλακισμένους να μεταφέρονται από το ένα αεροπλάνο σε λεωφορεία που έβγαιναν δηλαδή από αμερικανικά αεροπλάνα και έμπαιναν σε λεωφορεία. Υπήρξαν και κτίρια στο οποίο κρατήθηκαν, δεν ξέρουμε, μπορεί να ήταν 20 λεπτά, μπορεί να ήταν και 20 μέρες αναφέρθηκαν στα μέσα ενημέρωσης. Παρ' όλα αυτά δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι τώρα. Ελπίζω ότι μέσω της δικιάς μας έρευνας να πετύχουμε να φτάσουμε στην αλήθεια. Γιατί είμαι ένας από αυτούς που εδώ στο Κοινοβούλιο ...έχει δουλέψει για την ασφάλεια. Ναι, αλλά και στην ασφάλεια από την τρομοκρατία φυσικά. Αλλά εδώ αυτό, με αυτά τα γεγονότα υπονομεύουμε την ίδια μας την αξιοπιστία και δίνουμε επιχειρήματα στου, στις τρομοκρατικές οργανώσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γκόμες. Κυρία ευχαριστώ. Θα μιλήσω Ιταλικά. Είμαι πρόεδρος της Υποεπιτροπής ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ τη Λίμπε που οργάνωσε αυτή την ακρόαση σήμερα. Ελπίζω να καταφέρουμε να βρούμε κάποια στοιχεία, περισσότερες πληροφορίες και να υπάρξει διαφάνεια. Κυρία Χολ, είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εισαγάγει μια ε, διαδικασία λογοδοσίας σε περίπτωση παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, κάνετε αυτή την πρόταση Ευρωπαϊκές Αρχές. Τι απάντηση σας δώσανε. Επίσης είπατε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υποστηρίξουν την Επιτροπή ε, ΛΥΜΠΕ για να υπάρξουν ανεξάρτητες ε, έρευνες. Οι ευρωπαϊκές αρχές σε ποιο βαθμό σας βοήθησαν. Αυτά προς την κυρία φλότ. Κύριε Μπλακ τώρα. Είπατε ότι είναι σημαντικό να δούμε ότι υπήρχε ένα δίκτυο ολόκληρο. Με βάση τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, μάλλον προς αυτήν την κατεύθυνση και εμείς κινούμαστε, ότι υπήρχε δίκτυο. σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η ψηλά ιστάμενη πολιτική και στρατιωτική ήταν συνένοχη. Έπειτα, πέρα από την επιμελητία, χρειάζονται και κάποιες άδειε να δοθούν. Από τις αρχές. Άρα δόθηκαν άδειε από τις ευρωπαϊκές αρχές και φαντάζομαι ότι η Αμερικανική κυβέρνηση τη ζήτησε αυτές τις άδειε. Ξέρω ότι στη χώρα μου, τη Γερμανία, δημιουργήθηκε μια κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή που έδειξε ότι η αρχή συντονισμού ήταν ε, ένας υπουργός, ο οποίος ήξερε πάρα πολύ καλά τι γινότανε και έδωσε τις άδειε. Έχετε νέες πληροφορίες για αυτό το θέμα, κυρία Ίντβελ. Είπατε ότι η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη δεν έδωσε καμία σημασία στο θέμα αυτό. Όταν η Γερμανία ε, δημιούργησε αυτή την εξεταστική επιτροπή, τα εθνικά ΜΜΕ ενδιαφέρθηκαν για το θέμα αυτό και ενέκυψαν επί του ζητήματος. Αλλά όταν υπό αυτές τις συνθήκες δεν είναι δυνατόν ε, να έχει κανείς μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, που εμφανίζονται και προασπίζονται τις αρχές αυτές και υπάρχουν πολίτες οι οποίοι πέφτουν θύματα αυτών των κρατήσεων και μεταφορών. Ίσως θα έπρεπε οι πολιτικοί να βρουν καλύτερους τρόπους για να ελέγχουν καλύτερα αυτές τις κινήσεις διότι με το ε, την κάλυψη του απορρίπτου υπάρχουν κινήσεις οι οποίες δεν συνάδουν με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ κύριος Μικαέλσκι. Ευχαριστώ. Είμαι Πολωνός, αλλά θα προσπαθήσω να μιλήσω αγγλικά. θα, θα μιλήσω πολωνικά. Με συγχωρείτε, λάθος έκανα, ήθελα να πω ότι θα μιλήσω πολωνικά. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα τυπικό παράδειγμα μιας κατάστασης όπου αντιμετωπίζουμε ένα δίλημα. Ε, υπάρχει, πρέπει να υπάρχει ισορροπία ελευθερίας, ε, ασφαλείας ε, και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι η ελευθερία έχει λιγότερα δικαιώματα. Πρέπει να υπάρχει ένας ισοσκελισμός μεταξύ αυτών των ε, αρχών ε, και τα κράτη που συνέβαλαν εις ε, την εκστρατεία ε, στο Αφγανιστάν δεν το έπραξαν ε, γιατί ήθελαν να σκοτώσουν ή ήθελαν να ταξιδέψουν αλλά για να μπορέσουν να προλάβουν τρομοκρατικές επιθέσεις στο μέλλον. Τώρα βέβαια πρέπει να εξετάσουμε ε, έχοντας τη γνώση εκ των υστέρων ε, ε, ποιο είναι το κύρος ε, των ε, κινήσεων αυτών αλλά είναι μη, ένας πολύ σοβαρός αγώνας και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να πληρώσει και να επενδύσει εις ε, την ασφαλειά του οι, οι ψηφοφόροι μας δεν θέλουν να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες των χωρών και τα, τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε ζήσει με, υπό την προστασία των Αμερικανών. Είτε μας αρέσουν είτε όχι, πρέπει να αντιληφθούμε ότι... Ε, ε, βρισκόμαστε εκεί ε, διότι ε, μας το έχουν επιτρέψει οι Αμερικανοί πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε τους συμμάχους μας ή να αυξήσουμε πάρα πολύ τις αμυντικές μας δαπάνες ενώ οι ομιλητές μέχρι σήμερα δεν ήθελαν να επιλέξουν μεταξύ αυτών των δύο λύσεων δεν θέλουν ούτε να αυξήσουμε τις αμυντικές δαπάνες δαπάνες αλλά ούτε ε, να ε, ε, να συνεργαζόμαστε με τους Αμερικανούς. Επίσης στα ανθρώπινα δικαιώματα συνεργαζόμαστε ε, και έχουμε δικαίωμα να κρατήσουμε στα κράτη μας άτομα τα οποία θεωρούμε ότι ε, ε, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του κράτους μας χωρίς βέβαια να αποδεχόμαστε τους βασανισμούς. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Είτε παλεύουμε ε, για την ε, ασφάλειά μας ή ε, προσπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουμε δικαίωμα να μηνθούμε όχι όμως να βασανίσουμε και υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι ατυχώς έχουν διαπράξει αυτά τα, τα αδικήματα. Η κυρία Στίφλερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για το έγγραφο που μας δώσατε και θα αποτελέσει βάση των εργασιών μας. Πρέπει να σας πω ότι αντιθέτως με ό,τι ε, προεβλέπεται στο, συνημερίσια διάταξη προσπαθούμε εδώ ε, να αξιολογήσουμε την κατάσταση βάσει των νέων στοιχείων που προέκυψαν από το 2000 και καλό θα ήταν να έχουμε την άποψη ενός βουλευτή από τη Λιθιενία που συμμετείχε στην έρευνα αυτή που θα ήταν πολύ επικο, επικοδομητικό. Ξέρετε ότι το ΕΛΚ δεν είχε υπερψηφίσει την έκθεση και τα πορίσματα της προσωρινής επιτροπής και πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε πιο ε, σοβαρές αποδείξεις για να προβούμε σε σοβαρές ε, κατηγορίες αλλά από το 2007 έχουν προκύψει νέα στοιχεία πρέπει λοιπόν να υπάρξει επαναξιολόγηση θα ήθελα όμως να θέσω ερωτήματα στους ομιλητές δηλαδή πώς είναι δυνατόν να γνωρίζουμε συγκεκριμένα ότι ένας κρατούμενος μπήκε σε μία πτήση της CIA. Έχουμε φωτογραφίες, έχουμε έγγραφα, έχουμε ε, συγκεκριμένα στοιχεία στην περίπτωση του κυρίου Αμπουζαγιά. Πώς γνωρίζουμε ποια πτήση πήρε από την Ιορδανία ε, ε, μέχρι την Ευρώπη και είναι δεδομένο ότι με ορισμένα κράτη κράτη-μέρη έχουν συμβάλει ενεργητικά, τότε θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει μέτρα. Αλλά είμαι σκιώδης εισηγητής, θέλω να υπάρχει καλή συνεργασία με τους συναδέλφους, είτε εισηγητές είτε σκιώδης εισηγητές. Και σας ευχαριστώ. Η κυρία Φλότερ. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μπλακ. Όταν λέει ότι υπάρχουν προσγειώσεις αεροπλάνων σε αεροδρόμια χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχο συνόρων ή αστυνομικός. Τι θεωρεί ότι συνεπάγεται αυτό σαν ευθύνη της αλυσίδας διοικήσεως με ποιες, ποιους οργανισμούς των κρατών με ποιες υπηρεσίες, πόσο, ποιοι πρέπει να συμβάλλουν σε αυτή ε, την ενέργεια, διότι πολλές φορές ακούμε ότι υπάρχουν τόσες πληροφορίες εμπιστευτικές, απόρριτες, ε, διαβαθμισμένες που για να ρίξει φως κανείς σε αυτά τα θέματα είναι δύσκολο αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι και πολλά ε, στοιχεία τα οποία έχουν αποκαλυφθεί δεν έχουν χρησιμοποιηθεί χρησιμοποιηθεί και αντιτίθενται σε αυτή τη μέθοδο. Δηλαδή οι πληροφορίες αυτές που είναι απόρριτες ή εμπιστευτικές ή μη προσβάσιμες πόσο, πόσο κοινή συμφωνία και εκεί είναι η ευθύνη που είπε και η Σοφή Ιντβελτ ε, επιβάλλει αυτό ε, το νόμο της σιωπής μεταξύ κρατών και εδώ απευθύνομαι τους δύο προσκεκλισμένους δηλαδή είναι δυνατόν οι αρχές του ΝΑΤΟ να προβαίνουν σε τέτοιες διαβαθμίσεις ε, και σε τέτοιους χαρακτηρισμούς απορρίτων τέλος εάν υπάρχουν ε, ε, πληροφορίες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πώς Πού οφείλεται αυτό, στην ε, κακή θέληση αυτών που οργανώνουν ε, τις ε, έρευνες, προφανώς όχι όλους, αλλά υπάρχουν περιορισμένες εφαρμογές, οι εναλλασσόμενοι δεν το επιθυμούν, αλλά υπάρχουν εμπόδια και σύμφωνα με τις γνώσεις σας τι οδηγεί σε αυτά τα εμπόδια και ε, κάνω την ερώτηση σκεπτόμενη ότι θα ήθελα να μπορέσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να βρούμε τις ε, δυνατότητες να αναλάβουμε αυτή τη συλλογική ευθύνη και να αντιμετωπίσουμε αυτά τα εμπόδια. Πρέπει να είμαστε συνεκτικοί και θα πρέπει να μας εξηγήσετε πιο συγκεκριμένα ε, τι, πώς εσείς σχολιάζετε τη φύση αυτών των εμποδίων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ποτασιεβίτς ε, θα είστε ο τελευταίος ομιλητής προτού ακούσουμε τις απαντήσεις των ε, ε, συμμετεχόντων στη Σογγυλή Τράπεζα. Πολύ σύντομα, δεν έχω να κάνω σχόλιο, αλλά θα ήθελα να πω ότι εκτιμώ πολύ του εισηγητές ε, και την κοινοβουλευτική εργασία που έχει γίνει στο θέμα αυτό σχετικά με την παρουσία ε, και τις κρατήσεις από τη CIA στην Ευρώπη. Ε, ε, έχοντας δει πώς αντιμετωπίζουν οι διάφορες χώρες αυτή τη διαδικασία χωρίς να θέλω να υπερασπιστώ τον δημόσιο κατήγορο της ε, Πολωνίας πιστεύω ότι μετά από έτη ερευνών από, λέγεται από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα ότι ε, έχουν συμβάλει στις διαδικασίες αυτές και η υπεύθυνοι της Γενικής Εισαγγελίας της εποχής σημαίνει ότι οι εντολές αυτές έχουν εφαρμοστεί σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης. Το γεγονός ότι δεν παρίσταται ο Γενικός Εισαγγελέας ε, δεν, δεν αποτελεί στοιχείο κατεμέδια βασα το το γράμμα του μας λέγει ότι ούτως ή άλλως η διαδικασία ολοκληρώθηκε, δεν μπορεί να έρθει εδώ να μας αποκαλύψει ε, απόρριτα στοιχεία. Ε, αλλά ούτως ή άλλως ε, υπάρχει μία διαφορετική διαδικασία και ίσως η Πολωνική, το Πολωνικό Κοινοβούλιο ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία τουλάχιστον για να ολοκληρωθεί η έρευνα στην Πολωνία πιστεύοντας και ελπίζοντας ότι υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της Πολωνίας και άλλων χωρών οι οποίες ενδεχομένως βρίσκονται υπό την εξέταση της ιστορίας. Η κυρία Φαγιάν έχει ζητήσει το λόγο για πολύ λίγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Είναι σημαντικό το ότι ξεκίνησε αυτή η συζήτηση σήμερα, ε, έχοντας συγκεντρώσει τόσα στοιχεία, τόσα αποδεικτικά στοιχεία, έχοντας συζητήσει με τους Αμερικανούς ε, εμπειρογνώμονε με την ε, παρουσία των ΜΜΕ. Ε, εγώ δεν ήμουν τότε στο κοινοβούλιο της Επιτροπής ΒΑΒΑ, αλλά τότε ήμουν δημοσιογράφος στις Βρυξέλλες και θυμάμαι ότι η προσοχή των ΜΜΕ ήταν πολύ σημαντική στη δουλειά της προσωρινή επιτροπή του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ε, και πιστεύω το ίδιο θα γίνει και τώρα. Ε, με αυτή την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας, με αυτή την ακρόαση, με αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, πιστεύουμε ότι θα προσελκύσουμε την προσοχή των μέσων ενημέρωσης. Και αυτός είναι ένας τρόπος για να πιέσουμε πολιτικά τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αυτό είναι σημαντικό. Κύριε Μπλακ, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Αναφέρατε ότι ρωτήσατε 28 ευρωπαϊκές χώρες να συνεργαστούν και 14 χώρες αρνήθηκαν. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες ποιες χώρες αρνήθηκαν να συνεργαστούν. Γιατί για μένα, όταν λες όχι, έχεις κάτι να κρύψεις. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα συμφωνώ με κάποια από τα συμπεράσματά σας επίσης, ότι δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό να μιλάμε για ισχυρισμούς. Όταν έχουμε αποδεκτικά στοιχεία ότι η λιθουανική κυβέρνηση α, η ίδια αναγνώρισε την ύπαρξη δύο φυλακών, τότε για ποιους ισχυρισμούς μιλάμε. Μπορούμε να συζητήσουμε τότε τον τίτλο του εγγράφου μας για τους, α, τις φερόμενες μεταφορές και παράνο, υποτιθέμενες παράνομες κρατήσεις, οι καζόμενες. Ε, ας ακούσουμε λοιπόν τώρα τους ομιλητές. Η κυρία Χολ, θέλω να απαντήσω καταρχάς ε, στον Πολωνό Ευρωβουλευτή. Ε, είναι πολύ επίκαιρες αυτές οι κατηγορίες για την Πολωνία σήμερα. Ε, υπάρχει και ένα προηγούμενο μάλιστα. Έχουμε ε, καθόμαστε εδώ και λέμε, μιλάμε αρκετά κοινικά. Ε, στην ε, κοινοβουλευτική έκθεση του Λιθανικού Κοινοβουλίου υπάρχουν τρία άτομα που αναφέρονται. Και αυτές οι κατηγορίες ε, που βαραίνουν αυτά τα τρία άτομα θα αξιολογηθούν. Έγινε λοιπόν αυτή η έρευνα, αλλά έγινε μέσα σε κάθε μυστικότητα. Έχουμε ελάχιστες πληροφορίες, έκλεισε και θεωρήθηκε κρατικό μυστικό. Και αυτά τα τρία άτομα ποτέ δεν διώχθηκαν. Και όταν εμείς λέμε ότι επιφυλασσόμεθα να... και δεν αποφαινόμεθα, θέλουμε να δούμε τι θα προκύψει. Αυτό εννοούμε. Ε, γιατί έχουν ξαναγίνει τέτοια, έχουν ξαναγίνει προσπάθειε, αλλά τελικά δεν οδήγησαν πουθενά. Έχουμε απογοητευτεί στο παρελθόν, επομένω θέλουμε να δούμε κάτι παραπάνω. Για την ε, συνεργασία των ε, ευρωπαϊκών κυβερνήσεων ε, και το κατά πόσον ήταν συστηματική αυτή η φύση των επιχειρήσεων. Ε, θα πρέπει ε, στο άρθρο του European Voice να δείτε πώς, τι γλώσσα χρησιμοποιείται, τι φρασιολογία, όπου οι συντάκτες εκτιμούν την αμοιβαία αρρωγή που έχουν δώσει οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ε, πολύ ωραία. Υπάρχει συνεργασία ε, για θέματα καταπολέμησης της δημοκρατίας. Δεν έχουμε δει την ίδια συνεργασία α, στη δική μας την περίπτωση. Ωραία, όταν υπάρχουν διώξεις τρομοκρατών, όταν υπάρχει δίωξη της χρηματοδότησης της ε, τρομοκρατίας, υπάρχει αυτή η συνεργασία. Θα έπρεπε να υπάρχει αντίστοιχη συνεργασία για ε, τη διερεύνηση θεμάτων συνενοχής. Ε, τώρα, για αυτό που είπε η Γερμανίδα Ευρωβουλευτής, για το τι μπορείτε να κάνετε εσείς. Και μετά θα δώσω το λόγο στον Κρόφτον. Μην ξεχνάμε εγώ δεν θέλω να μιλήσω για να υπάρξει περισσότερη καθυστέρηση. Πρέπει να υπάρξει ε, λογοδοσία. Ε, πρόκειται για ένα παγκόσμιο σύστημα μεταφορών κρατουμένων, εμιστικών μυστικών ε, κέντρων κράτησης. Όταν δείτε, ας πούμε, την, τα Βαλκάνια, την Κεντρική Αμερική, τη Ρουάντα. εκεί μιλάμε για λογοδοσία. η λογοδοσία είναι ένα περίπλοκο θέμα και χρειάζεται χρόνο, ε, δύσκολες έρευνες. Ε. Αυτή η διαδικασία εδώ της ΛΥΜΠΕ είναι ακόμα ένα βήμα ε, στην όλη προσπάθεια. Δεν μπορώ να πούμε ότι χάσαμε τη μάχη για να χυθεί φως και να υπάρξει λογοδοσία. Πιστεύω ότι είμαστε στη δεύτερη φάση, το δεύτερο βήμα, σε μια προσπάθεια που μπορεί να πάρει και άλλα χρόνια, λίγο παραπάνω χρόνια. Απλώς πρέπει να δείτε το πλαίσιο και να δείτε και πού αλλού ε, απαιτείται λογοδοσία, αυτές τις χώρες που σας ανέφερα. Φυσικά η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη και κάθε κρατός μέλος που ε, φέρεται ως ε, συνένοχος σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να συνεργαστεί με την Επιτροπή ΛΥΠΕ. Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες. και είπα ότι η Φιλανδία θα έπρεπε να είχε δώσει το 2006 τα στοιχεία για τις απτήσεις αυτές. Ε, όταν ξεκίνησε αρχικά η προσπάθεια. Και άλλες ε, κυβερνήσεις έχουν στοιχεία και δεδομένα και θα έπρεπε να τους ε, γίνουν ερωτήσεις και θα πρέπει να τους ζητήσουμε να αποκαλύψουν αυτά τα στοιχεία. Αυτά τα, πράγματα μπορείτε να τα κάνετε εσείς, εδώ, οι ευρωβουλευτές. Κάτι άλλο που θέλω να πω. Ε, μίλησα με έναν υψηλό σκανδιναβό αξιωματούχο το Δεκέμβριο. Ε, και που με ρώτησε, «Ε, έγινε τίποτα. Ναι, κάτι έγινε, αλλά έχουμε αποδείξεις. Η υποχρέωση έρευνας είναι κάτι που φέρει το κράτος. Δεν την έχουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσει ε, δεν έρχονται εδώ πέρα με την απόδειξη, α πούμε, και το όνομα του, του δράστη. Αυτό που θέλουμε είναι να παίξει το ε, κράτος το ρόλο του, να χρησιμοποιήσει ε, όλους τους μηχανισμούς που έχει για να διερευνήσει όπως κάθε άλλο έγκλημα, όπως ερευνά κάθε άλλο έγκλημα. Ε, όπου πάμε ο Κρόφτον και εγώ, οι εισαγγελείς μας λένε ποιες είναι οι αποδείξεις σας. Η δουλειά τους είναι, των εισαγγελέων είναι να βρουν τις αποδείξεις, να ερευνήσουν με αυστηρότητα. Είναι δουλειά τους να βρουν το αποδεικτικό στοιχείο Κάποιοι αξιωματούχοι του Συμβουλίου της Ευρώπη είπαν ότι κάθε χώρα ε, για την οποία, την οποία βαραίνουν ε, οι τέτοιες χειρισμοί θα πρέπει να κάνει έρευνες ε, αυτών των τόπων εγκλήματος. Γιατί ας πούμε αυτές οι φυλακές, αυτές, η, μυστική χώρη κράτησης στη Λιθουανία είναι τόποι εγκλήματος. Και όταν υπάρχει έγκλημα, ένας εισαγγελέα δουλειά έχει να ερευνήσει. Τι κάνει με, τις, με τους τόπους εγκλήματος. Ε, τους ερευνά. Αυτό που ζητάμε από τα κράτη-μέλη ε, να κάνουν είναι να κάνουν τη δουλειά τους, να ερευνήσουν. Ευχαριστώ κυρία Χολ. Και τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Μπλακ που θα απαντήσει στις ερωτήσεις. Πολύ ωραία το θέσατε. Αυτό το θέμα των των αποδεικτικών στοιχείων, καθώς περνάει ο χρόνος και μου κάνουν αυτή την ερώτηση ξανά και ξανά, θεωρώ ότι δεν είναι η σωστή ερώτηση είναι πολιτική τακτική, ε, ούτω ώστε ε, ε, οι υπεύθυνοι να στρουφοκαμιλήσουν. Όπως είπε και η Τζούλια, θα έπρεπε ε, η σήμανση, θα έπρεπε ε, να, να κάνει τη δουλειά της, θα έπρεπε ο, ο ιατροδικαστής να κάνει τη δουλειά του στο Βουκουρέστι, στην Πολωνία. πότε, έγιναν, πότε έγινε η ερευνητική προσπάθεια, πότε πήραν δείγματα DNA, πότε ψάξανε τους τόπους εγκλήματος. Το, λέμε, το ονομάζουμε ε, πρόγραμμα μυστικών κρατήσεων. Δεν το λέμε τυχαία, γιατί ε, παρέκαμψε όλους τους ε, κλασικούς μηχανισμούς που, είχαν, ε, που έχουν δημιουργηθεί, ούτω ώστε ε, να ελέγχουμε, να ξέρουμε με ποιες συνθήκες κρατούνται φυλακ, ε, φυλακισμένοι κτλ. Εμείς δεν έχουμε τα στοιχεία να σας δείξουμε κάθε σκάλα, κάθε ε, που έχει σταματήσει, κάθε αεροπλάνο, ε, όλη τη διαδρομή, ε, έχουμε κάποιες ψηφίδες. Είναι ένα τόσο μεγάλο, εκτενές δίκτυο, τόσο πολλά τα στοιχεία, τόσο πολλά τα τεκμήρια. Αν έρθετε εδώ σε μένα και μου πείτε ότι υπάρχει έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων, τότε πείστε με για μια άλλη ιστορία, ότι κάτι άλλο συνέβη. Αλλιώς Έχουμε φτάσει σε ένα γελίο διέξοδο. Πολλές σωστές ερωτήσεις ε, ε, τέθηκαν ε, και ζητώ συγγνώμη των κροτέρων αν ξεχάσω να απαντήσω σε κάποια. Για, για την προσπάθεια ερωτήσεων που έκανε η Access for Europe. Δεν έχω φέρει αντίγραφο μαζί μου αλλά υπάρχει στο, στην ιστοσελίδα μας ε, και εκεί, στην ιστοσελίδα μας και, και εκεί υπάρχουν και τα στοιχεία των 14 χωρών. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα σε αυτές τις χώρες. Σε αυτή την έκθεση ήρθαμε σε επαφή και με το Eurocontrol, που αρνήθηκε να μας δώσει πληροφορίες, γιατί είπαν ότι είχαν μια πολιτική μη αποκάλυψης τέτοιου είδους πληροφοριών σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ε, νομίζω όμω ότι θα τι έδινε αυτέ τι πληροφορίε στο Κοινοβούλιο. Και ακριβώ γι' αυτό το Κοινοβούλιο είναι πολύτιμο όργανο. Μπορεί να παίξει αυτό το πολύ σημαντικό ρόλο ε, και μπορούμε, ε, χάρη στην παρέμβαση του Κοινοβουλίου, να διευρύνουμε τι πληροφορίε που έχουμε στη διάθεσή μα. Άλλε ερωτήσει. Για τη συνενοχή των πολιτικών ε, σε διάφορες χώρες δεν είναι οι πληροφορίες που εγώ έχω στη διάθεσή μου, που φτάνουν σε μένα. Ε, εγώ ε, βρίσκω άλλου τύπου στοιχεία. Αλλά στην ε, λιθουανική έρευνα αυτό προκύπτει ότι υπάρχει τέτοια συνενοχή. Επίσης, δεν απόκειται σε μένα να υποδείξω τι μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο στα πλαίσια της εντολής του. Ένα καλό σημείο αφετηρίας θα ήταν να αναγνωρίσει ότι παρότι Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, κάποιες αμφισημίες. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου ο όρος ισχυρισμός ε, δεν έχει νόημα. Ισχυρισμοί. Ούτως ή άλλως ε, και οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, έχουν παραδεχτεί ότι υπήρχε αυτό το πρόγραμμα, ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν το παραδέχονται ότι έγινε. Αυτό είναι το θέμα. Νομίζω ότι αυτά είχα να πω. Και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να μου στείλετε email, να μου υποβάλλετε κάποιες άλλες ερωτήσεις. Αν θεωρείτε ότι δεν έχω απαντήσει επαρκώς ε, στο ερώτημά σας, ε, μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μου. Κύριε Χολ, θέλετε κάτι να προσθέσετε από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ναι, πολύ σύντομα. Για το θέμα των μυστικών ε, υπηρεσιών, οι βουλευτές πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν να αλλάξει κάτι, γιατί είναι το τελευταίο όριο που λείπει η διαφάνεια και η δημοκρατία. Συναντιόμαστε με υψηλό επίπεδο πολιτικούς και ορισμένοι μας λένε «Καλή την πίστη». Δεν είμαστε σίγουροι. Δεν λέω ότι είναι πολλοί, αλλά υπάρχουν κάποιοι. Μιλούν ανοιχτά για διαφορετική συχνότητας επικοινωνία. Δεν πρόκειται μόνο για τη συχνότητα που είναι η πολιτική, υπάρχουν πολλών επιπέδων συχνότητες. Γι' αυτό μιλάμε για δίκτυο. Βλέπετε διαφορετικοί ε, παράγοντες ε, δρούν σε διαφορετική συχνότητα. Αυτό που είναι λοιπόν σημαντικό όσο προχωράμε είναι το κάθε επίπεδο να αναθεωρήσει τη δημοκρατική, το δημοκρατικό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Το είδαμε και ε, με την έκθεση ΦΑΒΑ και φτάσαμε και μέχρι τις εκδόσεις στη Συρία. Συνεπώς πρέπει να υπάρξουν συστάσεις για να υπάρξει αλλαγή ε, σε αυτό που είναι αντίστοιχα η CIA και το FBI. Πρέπει να δούμε ποια είναι τα στοιχεία που έχουμε, τι ξέρουμε για τα θύματα και να φροντίσουμε να μην ξανασυμβούν τέτοια πράγματα σε ευρωπαϊκή επικράτεια. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ και την κυρία Χόλ και τον κύριο Μπλακ και όλους τους ευρωβουλευτές για όσα μας είπανε. Η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Έχουμε όμως καθυστερήσει λίγο, γι' αυτό ας περάσουμε αμέσως στο δεύτερο κομμάτι της ακρόασής μας, που είναι παρουσίαση συγκεκριμένων περιπτώσεων. Ο κύριος Τζον Γκότς δεν ε, μπόρεσε να έρθει, έχει ενεργημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις ε, πρόκειται για δημοσιογραφικές έρευνες του Εθνικού Γερμανικού Τηλεοπτικού Σταθμού ΑΕΡΔΕ σχετικά με το μυστικό κέντρο κράτηση τη CIA στην Ρουμανία. Η κυρία Μάντα Τζάκοψον όμω είναι εδώ, που είναι δικηγόρο του Αμπού Ζουμπαϊντάχ, που είναι θύμα παράνομη κράτηση τη CIA στην Ευρώπη. Η κυρία Μάντα Τζάκοψον λοιπόν θα πάρει τώρα το λόγο θα μας ε, κάνει τη δικιά της παρουσίαση και μετά θα στραφούμε στο δεύτερο προσκεκλημένο μας που είναι ο Άνταμ Μποντνάρ και τέλος ε, θα ακούσουμε την κυρία Άμριτ Σινγκ. Καλώς ήρθατε όλοι. Παρακαλώ. Προχωρήστε γρήγορα και τελειώ θα μείνουμε πίσω στο χρόνο. Παρακαλώ κύριε Τζάκοψεν. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Ονομάζομαι Αμάντα Τζάκοψεν, είμαι Αμερικανίδα, δικηγόρος και εκπροσωπώ το φυλακισμένο στο Γουατάνομο και τέο θύμα παράνομης κράτησης της CIA, τον Αμπού Ζουμπαντά. Είναι γνωστό με αυτό το όνομα και το ολόκληρο όνομά του είναι Ζάιν Αμπιντήρ Μουχάμετ Χουσίν. Ε, τον εκπροσωπώ από τότε που έφτασε στο Γουατάνομο μετά από παράνομη κράτηση της ε, CIA και του δόθηκε το δικαίωμα να έχει δικηγόρο. Η κράτησή του θεωρώ ότι εξακολουθεί να είναι παράνομη και προσπαθώ να το αποδείξω αυτό όπως επίσης να τον υποστηρίξω και για άλλα θέματα όπως η παράνομη κράτησή του από τη CIA στην Ευρώπη. Τον έχω επισκεφθεί στο Guantanamo Bay κάθε μερικούς μήνες, πηγαίνω τα τελευταία χρόνια. Σήμερα βρίσκομαι εδώ για να σας μιλήσω εκ μέρους του. Δηλαδή, σήμερα βρίσκομαι εδώ για να μιλήσω εκ μέρους ενός θύματος τέτοιας παράνομης κράτησης στα πλαίσια του προγράμματος του σχετικού της CIA. Ξέρω ότι δεν είναι πολλοί που έχουν την ευκαιρία αυτή. Να ξέρετε ότι έχοντας μιλήσει μαζί του, τον έχω γνωρίσει και ως προσωπικότητα και για την ε, κατάστασή του. Βέβαια, τόσο εγώ γνωρίζω κανονικά είναι απόρριτα. Ελάχιστα πράγματα μπορώ να πω εδώ δημόσια. Το ερώτημα που θέτεται σήμερα είναι τι Νέες εξελίξεις έχουμε όσον αφορά την, την εικαζόμενη παράνομη κράτηση και μεταφορά κρατουμένων στην Ευρώπη από τη CIA. Ε, λοιπόν, όσον αφορά τον πελάτη μου, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Περνούν τα χρόνια, δεν υπάρχει λογοδοσία και κάθε τόσο ε, συναντάω στο κελί απομόνωσης τον πελάτη μου. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα επειδή φαίνεται ε, ο κόσμος συνειδητοθεί όλο και περισσότερο ότι ο χρόνος έχει περάσει. Ε, δεν ασχολείται κανείς με το θέμα αυτό, δεν το θεωρεί πια επίγον και ούτε ασχολείται με την αδικία που γίνεται σε όλα αυτά τα θύματα. Για τον πελάτη μου όμως η αδικία αυτή συνεχίζεται και πρέπει να υπάρξει λογοδοσία. Υπάρχει ανάγκη για λογοδοσία. Όπως είπε και ο κύριος Μπλακ πριν, Αύριο 28 Μαρτίου 2012 έχουμε ακριβώς 10 χρόνια, μια δεκαετία δηλαδή από τότε που κρατείται ο πελάτης μου. Και ο κόσμος εκπλήσεται μερικές φορές που μαθαίνει ότι 10 χρόνια και στα 10 χρόνια αυτά δεν έχει υπάρξει απαγγελία κατηγορία σε βάρος του πελάτη μου. Δεν ε, είπε κανένα δικαστήριο ότι έπρεπε να βρίσκεται στη φυλακή. Το 2002 όταν συνελήφθη ο πελάτης μου και πέρασε από διάφορες μυστικές ε, φυλακές, η ψηλά ειστάμενη εξωματούχη των ΗΠΑ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημόσια είπαν ότι ο πολίτης μου ήταν ε, το νούμερο 3 στην Αλκαΐδα. Υπεύθυνο για διάφορε δραστηριότητε, διευκόλυνσε διάφορε εγκληματικέ ενέργειε, συνεργάστηκε με τον Πιλάτη κτλ. Ότι συμμετείχε προσωπικά σε επιθέσει τη 11η Σεπτεμβρίου και σε όλες τις μεγάλες δραστηριότητες της ε, Αλκαΐντα και τη γνωρίζει, γνώριζε τα μελλοντικά σχέδια της Αλκαΐντα. Όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί όμως είναι ψευδείς γιατί ο Μπού Ζουνταϊντά δεν ήταν μέλος καν της Αλκαΐντα, πόσο μάλλον το νούμερο 3. Δεν συμμετείχε ούτε στο σχεδιασμό ούτε στην εκτέλεση επιθέσεων της Αλκαΐντα. Δεν ήταν δηλαδή αυτό που η κυβέρνηση υποστήριζε ότι ήταν. Μπορεί να εκπλήσει αυτό, αλλά η Αμερικανική κυβέρνηση είπε ότι δεν υποστηρίζει πλέον τους ισχυρισμού αυτού σε βάρος του πελάτη μου. Υπήρξαν δύο έρευνες που έγιναν όσο αφορά την μεταχείριση του πελάτη μου στη Λιθουανία και στην Πολωνία. Πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο της Λιθουανίας και το πρόγραμμα της CIA e ξεκίνησαν από τον Αύγουστο του 2009, τότε δηλαδή άρχισαν τα πράγματα να γίνονται γνωστά. Τον Ιανουάριο του 2011 υπήρξε έρευνα για τους ισχυρισμούς αυτούς από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Λιθουανίας για την Εθνική Ασφάλεια και την Άμυνα και κατέληξε στο ότι η CIA ε, όντως είχε αεροπλάνα στη Λιθουανία. Επίσης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Λιθουανία πήρε, έλαβε έτοιμα να φιλοξενήσει κρατούμενους και να προσφέρει ε, διευκολύνσεις τις οποίες και έφτιαξε στο μεταξύ. Άρα λοιπόν πρόκειται για άτομα όπως ο πελάτης μου που όντω βρέθηκαν στην Λιθουανία. Μετά σταμάτησε η έρευνα. Χωρίς να το ψάξει περισσότερο η έρευνα, σταμάτησε απλώς. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν μπορούσαν να γίνουν πλέον έρευνες πάνω σε αυτήν την υπόθεση. Ακούσαμε και από τη Διεθνή Εμνηστία ότι υπάρχουν ε, αποδείξεις για το ότι ο πελάτης μου, για παράδειγμα, μυστικά κρατεί σε φυλακή στη Λιθουανία. Όμως η λιθουανική κυβέρνηση δεν δέχτηκε τις αποδείξεις ε, αυτές και αρνήθηκε να ξανανοίξει την έρευνα. Εκ μέρους λοιπόν του Ναμπού Ζιβετάια και εγώ και ο πελάτης μου ζητούμε, ε, κάναμε μάλλον προσφυγή στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο και τα όσα έγιναν στη Λιθουανία. Τώρα, όσον αφορά την Πολωνία, ενώ από το 2005 υπάρχουν στοιχεία για μυστικές φυλακές στη χώρα, η έρευνα ξεκίνησε μόνο το 2008. Τώρα που είμαστε στο 2012, η έρευνα δεν έχει καταλήξει ακόμα σε συμπεράσματα. Και μάλιστα τον προηγούμενο μήνα έφυγε από την εισαγγελία της Βαρσοβίας υπόθεση και πήγε μετάδες χιλιόμετρα μακριά στην Καρκοβία. Η αλλαγή αυτή να φύγει δηλαδή από τα χέρια κάποιου ανθρώπου που ήταν εξοικειωμένο με την υπόθεση και να πάει στα χέρια κάποιου άλλου που δεν την γνωρίζει, σημαίνει ότι θα καθυστερήσει ακόμα περισσότερο η έρευνα. Και παρά το ότι και τα μέσα ε, ενημέρωση και ο ίδιο ο πελάτη μου ζητήσαν εξηγήσει, δεν πήρανε καμία γιατί έγινε αυτή η αλλαγή. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Στα πλαίσια μιας έρευνας το 2011 ο επικεφαλής εισαγγελέα ε, ε τα καθήκοντά του και ανέλαβε άλλες υποθέσεις. Υπάρχουν λοιπόν τέτοια εμπόδια και καθυστερήσεις. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και στην περίπτωση του πελάτη μου, ο οποίο και πάλι προσφεύγει στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και για αυτή την υπόθεση τη Πολωνία. Παρά το γεγονό λοιπόν ότι η έρευνα δεν γίνεται καλά, ε, εκτό από τι καθυστερήσει και τι αλλαγέ αυτέ υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Το πρώτο έχει να κάνει με την πρόσβαση του πελάτη μου στην έρευνα. Διότι γνωρίζουμε από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο ότι υπάρχει υποχρέωση στα πλαίσια μιας ε, έρευνας. Ε, υπάρχει λοιπόν υποχρέωση να ενημερώνεται και ο πελάτης, να του προσφέρεται η πρόσβαση στις πληροφορίες. Εδώ πρόκειται για ένα θύμα, ένα θύμα το οποίο δεν μπορεί εφόσον δεν γνωρίζει ε, τα στοιχεία που υπάρχουν γύρω από την υπόθεση να βοηθήσει. Το 2010 ο Μπούζου Δεντά ε, πήρε το καθεστώς του θύματος του παραχωρήθηκε αυτό το καθεστώς. Όμως ούτε ο πελάτης μου, ούτε εγώ, ούτε ο Πολωνός ο δικηγόρος του είχαν πρόσβαση στην έρευνα. Στην Πολωνία ο δικηγόρος μου, Τσακόσκι, ζήτησε πρόσβαση στην έρευνα. Ο ίδιος δεν έχει όμως πρόσβαση στην υπόθεση αυτή, όπως δεν έχω κι εγώ. Σήμερα, λοιπόν, ο κύριος Σαλκάσκι μπόρεσε να δει μέρος μόνο των στοιχείων που υπάρχουν για την υπόθεση αυτή στην Πολωνία. Τα υπόλοιπα ότι είπαν δεν τον αφορούν είναι απόρριτα. Ο Πολωνός δικηγόρος λοιπόν μπόρεσε να δει ένα τμήμα του φακέλου. Αυτό το, αυτό το τμήμα όμως είναι ένα μικρό και ακόμα και από αυτό που θα μπορούσε να δει, ε, δεν έχει καταφέρει να έχει πρόσβαση σε ολόκληρο αυτό το κομμάτι. Θέλουν να οριστεί η ημερομηνία και ορίστηκε, αλλά πριν φτάσει η ημερομηνία αυτή, ο φάκελος μεταφέρθηκε από τη Βαρσοβία στην Κρακοβία, οπότε πάλι υπήρξε καθυστέρηση. Ο κύριος Κατάρσκη τελικά είδε ένα κομμάτι και θα έλεγα ότι το κομμάτι αυτό δεν έχει και πολύ νόημα. Δεν έχει πρόσβαση εξάλλου ούτε σε υπολογιστή για να μπορεί να το χρησιμοποιήσει, για να συνδέσει τα στοιχεία, για να μπορεί να συγκεντρώσει κάτι. Δηλαδή δεν του επιτρέπουν να γράψει τίποτα από τα όσα υπάρχουν στον ε, φάκελο και όμως υπάρχουν χιλιάδες σελίδες και δεν μπορεί να σημειώσει τίποτα. Γιατί περνάει από την ασφάλεια και δεν μπορεί να έχει απάνω του κανένα σημείωμα σε σχέση με τα όσα συμβουλεύτηκε και με τα έγγραφα που είδε. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Θεωρείται ότι παραβιάζει τον νόμο αν σημειώσει κάτι από τα στοιχεία στο οποίο έχει πρόσβαση. Και αυτό όπως εμποδίζει την ε, τον πελάτη Επίσης δεν μπορεί να μιλήσει για την ουσία των πληροφοριών που θα έχει διαβάσει στο φάκελο. Παρά μόνο σε που και αυτοί έχουν δικαίωμα πρόσβαση στο φάκελο αυτό. Άρα ούτε με τον Αμπουζουμπάντα. Ενώ είναι θύμα, τελικά του επέτρεψαν να δει τα ίδια στοιχεία που μπορεί να δει και ο δικηγόρος. Και τελικά ακριβώ επειδή κρίθηκε θύμα ο κύριος ε, Σουμπαντά, μπορεί και ο δικηγόρος του να έχει πρόσβαση στο φάκελο αυτό. Παρόλα αυτά, ο πελάτη μου εξακολουθεί να είναι στη φυλακή στο Γουαντάναμο. Δεν μπορεί να πάει στην Πολωνία να συμβουλευτεί το φάκελο. Και άρα, ενώ θα είχε δικαίωμα να το συμβουλευτεί, δεν τον έχει συμβουλευτεί και άρα ο δικηγόρο του δεν μπορεί να μοιραστεί μαζί του στοιχεία τα οποία έχει διαβάσει το φάκελό του. Και στην περίπτωση του Μπουμαχάμετ και του Σουκαμάν, το Ηνωμένο Βασίλειο έστειλε απόρριτο φάκελο στο Γουαντάναμο για να μπορέσουν οι κρατούμενοι αυτοί να ενημερωθούν. Στην περίπτωση του πελάτη μου δεν έχει γίνει αυτό, ενώ θα μπορούσε να γίνει. Είναι κάτι το οποίο ζητούμε προκειμένου να μπορέσει και ο πελάτης να ενημερωθεί για όσα τον αφορούν. Ένα άλλο θέμα που προκύπτει όσον αφορά την έρευνα στην Πολωνία είναι ότι δεν υπάρχει διαφάνεια. Η υποχρέωση ενημέρωσης προς το θύμα και να μπορεί να αντιδράσει στις πληροφορίες αυτές στο θύμα είναι κάτι που αποτελεί υποχρέωση σύμφωνα με το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου. Πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Όμως ε, στο κομμάτι στο οποίο έχει πρόσβαση ο Πολωνός δικηγόρος, ο κύριος Κοτσάσκι, λέει ότι τίποτα δεν έχει δει, τίποτα προς το παρόν που πραγματικά να πρέπει να τηρηθεί απόρριτο. Ό,τι έχει δει είναι θέματα που μπορούν ε, κάλλιστα να είναι δημόσια. Δεν υπάρχει λόγος για απόρριτο. Άρα το καθεστώς του απορρίτου αποδεικνύεται ε, περιττό. Ο κύριος Ζεκάρσκι ζητάει να μην είναι πλέον απόρριτα τα στοιχεία αυτά και σύμφωνα με τον δικηγόρο αυτό δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίσει τη διακατάσταση. Δυστυχώς πολλά πράγματα μένουν κρυφά από τον κόσμο, από το κοινό. Υπάρχει και θέμα γνωμοδότησης, νομικής γνωμοδότησης όσον αφορά την ε, κατάσταση των ε, ε, παράνομων κρατήσεων. Η νομική αυτή γνωμοδότηση είναι ένα έγγραφο το οποίο θα μπορούσε να κυκλοφορήσει. Όμως δεν γίνεται αυτό. Θα ήταν καλύτερο έστω και μια περίληψη να υπάρχει κάποια διαφάνεια τουλάχιστον. Το τελευταίο πρόβλημα σχετικά με την έρευνα. Ο Αμπού Σουμπαντά και ο δικηγόρος του ξέρουν ότι υπάρχουν αρκετές πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί για να ληφθεί κάποια απόφαση. Όμως η εισαγγελία δεν έχει απαγγέλει κατηγορία ακόμα. Οι διαδικασίες, σύμφωνα με τον κύριο Ζεγάσκη, έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο που δεν υπάρχει πια πολύ περιθώριο, πρέπει να πάρθει κάποια απόφαση. Μετά τη δουλειά που έκανε ο εισαγγελέα πάντως, τέσσερα χρόνια έρευνας από το 2008 μέχρι το 2012, Τώρα λοιπόν, μετά από αυτά τα τέσσερα χρόνια, έφυγε από τα χέρια του φάκελο και πήγε στην Κρακοβία, όπω σα είπα. Πριν ξεκινήσει η ακρόαση αυτή, σήμερα το πρωί ακούσαμε ότι τον Ιανουάριο πριν γίνει η μεταφορά στην Κρακοβία ε, κατηγορήθηκε ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Και παρά το γεγονός ότι η πολωνική κυβέρνηση ε, μπορεί να πει ότι δεν υπάρχει συνεργασία από τις Αμερικανικές αρχές, παρόλα αυτά ο κύριος Τσακαβάσκη λέει ότι θα μπορούσε να βγει κάποια απόφαση παρόλα αυτά βάσει των πληροφοριών αυτών. Ζητάω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει έκκληση στι κυβερνήσει τόσο τη Πολωνία όσο και τη Λιθουανία να πιέσουν ώστε να ληφθούν οι δύσκολε αποφάσει που πρέπει να ληφθούν τώρα. Σα ζητώ να κάνετε έκκληση στις χώρες αυτές να προσφέρουν πρόσβαση στα στοιχεία για τον πελάτη μου, ώστε να μπορέσει να ενημερωθεί και ε, ο πελάτης μου και ο Πολωνός δικηγόρος του και εγώ. Επιπλέον, ζητώ από τις κυβερνήσεις αυτές να μην κρατούν απόρριτες όλες αυτές τις προφορίες να ενημερώνουν περισσότερο τον κόσμο. Παρά την κακή μεταχείριση που υπέστη 10 χρόνια ο πελάτης μου, δεν ζητάει αποζομίωση, ζητάει μόνο δικαιοσύνη. Να μάθει ο κόσμος ποιος είναι πραγματικά και ποιος δεν είναι. Γιατί ο κόσμος νοιάζεται για το τι γίνεται μυστικά από τις κυβερνήσεις και δεν ε, θέλουν να είναι οι χώρες τους υπεύθυνε για τέτοια μεταχείριση. Αυτά είναι σημαντικά για τον ε, πελάτη μου, αλλά και για το κράτος δικαίου, γιατί αν δεν απαιτήσουμε λογοδεσία από αυτούς οι οποίοι παραβιάζουν τον νόμο, είναι σίγουρο ότι τέτοια πράγματα θα ξανασυμβούν. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι ερωτήσεις έχετε. Ευχαριστώ την κυρία Γιάκοψον για την ε, παρουσίασή της και τώρα... Θα ήθελα να ακούσω τον ε, κύριο Άνταμ Μπότνερ, αντιπρόεδρο του Helsinki Foundation for Human Rights, σχετικά με την κατάσταση στην Πολωνία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ. Έχω μία πολύ σύντομη παρουσίαση για να παρουσίασω ορισμένα στοιχεία της ομιλίας μου. Εκπροσωπώ μία οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Πολωνία και έχουμε εμπλακεί στην Πολωνία από την αρχή και προηγουμένως ο καθηγητής Άντριου Ζαμπίνσκι ήταν υπεύθυνο ε, και στη συνέχεια εγώ ενέλαβα την, ε, την διεύθυνση αυτής της ε, υποθέσεως ε, είναι προφανές από την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η πολιτική ακολουθεί ε, μία ε, ότι η Πολωνία ακολουθεί μία πολιτική πλήρης απορρίψεως και αρνήσεως ότι υπήρξαν πτήσεις ή αφήξεις σε συγκεκριμένα σημεία. Πρέπει να σας πω ότι ο υπεύθυνος Πολωνία που έφερε το θέμα αυτό προς ο κύριος ε, Ιούζεφ ε, ε, Πάνερ και ήταν ο μόνος θαραλέος Πολωνός ο οποίος θεώρησε ότι έπρεπε το θέμα αυτό να εξηγηθεί και να του δοθεί ιδέουσα προσοχή και δημοσιότητα. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα τώρα στην Πολωνία, διότι όπως είπε και ο Ντίκ ε, βλέπουμε ότι υπάρχει μία δυναμική για την αλήθεια. Δηλαδή υπάρχουν όλο και περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες, δημόσια, που, θεωρούν, που καθιστούν πολύ πιθανόν ότι υπήρξαν φυλακές της CIA στην Πολωνία και ξεκινώ καταρχήν με την παρουσίαση της οργάνωσής μου ε, και ε, πρέπει να σας πω ότι από το 2007 και εντεύθεν έχουμε ε, ζητήσει πληροφορίες από τις αρχές της Πολωνίας και στη συνέχεια μας ε, έδωσαν ανεπίσημα πληροφορίες ε, οι αρχές παρακολουθήσεως της σεναρίου κυκλοφορίας ότι υπήρξαν ανεπίσημες αφήξεις αεροπλάνων εις τα αεροδρόμια της Πολωνίας στην εποχή που το Κοινοβούλιο και άλλες αρχές δεν είχαν καμία ε, ε, επίσημη επιβεβαίωση από τις πολωνικές αρχές. Άρα τα στοιχεία αυτά απέδειξαν ότι υπήρχε ε, συνενοχή εις αυτής της πτήσης ε, μεταξύ του 2002 και το Δεκέμβριο του 2003 και το 2010 μας ε, ειδοποίησαν από τις αρχές των συνόρων ότι είχαν υπάρξει άδειες συνοριακές για την άφηξη αυτών των, πλή, των αεροπλάνων και για τα αεροπλάνα και για τα πληρώματά τους πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι υπήρχαν στα αεροπλάνα αυτά και ε, επιβάτες που έφθαναν αλλά και πτήσεις που ανεχώρησαν χωρίς επιβάτες. Το 2003 όμως έφτασε ένα αεροπλάνο χωρίς επιβάτες και έφυγε με πέντε επιβάτες και αυτό συμπίπτει με το κλείσιμο της εγκαταστάσεως του, της CIA στην Πολωνία. Ο Άνταμ Σιρκόσκι που είναι γνωστός από το, την τηλεοπτική εκπομπή Πανοράμα έχει επιβεβαιώσει τα στοιχεία αυτά τα οποία και εμείς συλλέξαμε. Το 2008 όπως σας είπα και προηγουμένως ξεκίνησε επίσημα η έρευνα. Πρέπει λοιπόν να τονίσω ότι για τρία χρόνια δεν υπήρξε μια έρευνα. Η πρώτη ε, επίσημη αναφορά εις ε, τα κέντρα αυτά ε, ήταν το 2005 μέχρι το 7 δεν έγινε τίποτα ξεκίνησε η επίσημη έρευνα το 2008 και πέρασε από διάφορες φάσεις. Καταρχήν και αυτό νομίζω είναι πιο σημαντικό για την ακρόαση αυτή ε, ήταν ότι οι ανακριτές απεμακρύνθησαν ε, από ε, την περίπτωση αυτή χωρίς καμία αιτιολογία. Ο κ. Ζεκνεύσκη το 2011 χωρίς καμία εξήγηση. Και επίσης πολύ πρόσφατα το Φεβρουάριο του 2012 ένας άλλος ανακριτής, ο κ. Βάλτε Μαρτέ, απεμακρίνθη απεμακρύνθη ε, και μεταφέρθηκε από την εισαγγελία της Βαρσοβίας στην εισαγγελία της Κρακοβίας όπου βρίσκεται τώρα και θα σας πω στη συνέχεια πώς το εξηγώ. Ε, επίσης σημαντικές πληροφορίες <coughs> που αναφέρονται στις έρευνες στην Πολωνία ε, μας δείχνουν ότι δύο άτομα έλαβαν καθεστώς θυμάτων στην Πολωνία, ε, δηλαδή υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι είχαν κρατηθεί στην πολωνική επικράτεια ε, πρόκειται για τον κύριο Ανασύρη και δεύτερον για τον Απού Ζουμπάιμπτα, ε, τους δύο τους οποίους ακούσατε και προηγουμένως οπότε έχουν ένα επίσημη αναγνώριση επισήμου καθεστώτος ε, σαν θύματα έχουν νομική κάλυψη από Πολωνούς δικηγόρους που μπορούν να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες για την υπεράσπισή τους. Ε, υπάρχει επίσης και δικηγόρος ε, ε, για τον Βάλι Μπιν νατά στην Αμερική, ο οποίος είχε κρατηθεί στο Γκουαντάναμο, αλλά μέχρι στιγμής από ό,τι ξέρω δεν έχει αναλάβει επίσημα δράση ή κάποια διαβήματα και έχουν ζητηθεί πληροφορίες ε, κατόπιν των οποίων έχουν επιτύχει η ενημέρωση από τις πολωνικές αρχές σχετικά με τις έρευνες και οι έρευνες αυτές αναφέρονται εις ε, ε, την κατάχρηση της δυνάμεως των επισήμων και οδήγησε σε συνεργασία με την CIA ε, και ε, ε, σε άτομα σχετικά με τη CIA. Επίσης ζητήθηκε ε, νομική βοήθεια κατά τρόπον ώστε να ε, εξεταστούν ορισμένοι μάρτυρες οι οποίοι βρίσκονται στην Αμερικανική επικράτεια αλλά η πρώτη τέτοια αίτηση απερίφθηκε από τη ΣΥΠΑ και στην δεύτερη αίτηση ούτε καν υπήρξε απάντηση οπότε δεν υπάρχει καμία συμμετοχή και συνεργασία με τις Αμερικανικές Αρχές σχετικά με αυτές τις διαδικασίες και έρευνες. Έχουν αναλυφθεί ορισμένα διαδικαστικά ε, διαδικαστικές ενέργειες, δηλαδή ακροάσεις μαρτύρων χωρίς να ξέρουμε αν έχουν εξαιρεθεί από το σύστημα του κρατικού απορρίτου και δεν έχουμε στοιχεία σχετικά με αυτές τις ε, εξετάσεις μαρτύρων. Και τέλος θα ήθελα να σας πω ότι όσον αφορά την ε, έρευνα υπάρχουν και άλλα βασικά γεγονότα πρόσφατα και ε, υπήρξε ε, μία δήλωση του άντρε Σέρεμετ στο στη γερουσία της Πολωνίας προς τον Ιούζεφ Πίνορο ο οποίος είναι ένας Πολωνός πολιτικός και είχε ερωτήσει ε, πού βρίσκεται η εξέταση σχετικά με το θέμα αυτό, τι θα συμβεί. Δεν υπήρξαν επίσημα στοιχεία απάντησης, αλλά ελέγχθη ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και ε, αυτός συνέκρινε τη σημασία αυτής ε, της ε, ε, της ανακρίσεως με την εξέταση του πολωνικού αεροπορικού δυστυχήματος όπου υπήρξαν τόσα επιφανή θύματα και ε, τελικά ε, έχει εξαιρεθεί ο πρώην πρόεδρος Αλεξάνδρε Δεφεσνιέσχη της Πολωνίας από το καθεστώς κρατικού απορρίτου και ο κύριος Κομορόφσκι ε, αρνήθηκε να άρει το απόρριτο για αυτόν τον πρώην πρόεδρο ο οποίος δεν μπορεί να εξεταστεί Εξού και ε, στο ε, Δικαστήριο ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ξεκίνησε μία ενέργεια κατά της Πολωνίας σε σχέση με αυτές τις κινήσεις της CIA βάσει του άρθρου 2 και 3 του ανθρωπιστικού κώδικα που υποχρεώνει να εξεταστούν ορισμένες συνθήκες για ενδεχόμενη συνεχιζόμενους βασανισμούς και κακομεταχειρήσεις στην πολωνική επικράτεια και ε, έκδοση ε, προς ε, τις Ηνωμένε Πολιτείες, πράγμα το οποίο έγινε στην περίπτωση του κυρίου Αλνασίρη. Για την έκθεση αυτή μου επιτράπει επίσης να σας πω και αυτό μου το επέτρεψε ο κύριος Τόμας Χάμεμπεργκ που είναι ο σύμβουλος του ε, Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρωπίνα δικαιώματα ε, να, ε, ο οποίος προσπαθεί να πείσει τις πολωνικές αρχές ότι η περίπτωση είναι πολύ σοβαρή και το 1911 με κάλεσε ή το Στρασβούργο, στο γραφείο του μαζί με αυτούς οι οποίοι χειρίζονται την υπόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτή και ε, μου παρουσίασε όλα τα στοιχεία τα οποία διαθέτει. Ουσιαστικά μου έδωσε δηλαδή λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη φυλακών της CIA στην Πολωνία. Δεν ξέρω όμως τι έχει γίνει με το υλικό αυτό. Ελπίζω ότι έχει περιληφθεί στην δικογραφία της περιπτώσεως και θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο. Ε, τέλος, στις ε, αρχές Μαρτίου 2012 σε μία πολωνική εφημερίδα ε, δημοσιεύτηκε ένα άρθρο σχετικά με τις κατηγορίες για φυλακές της CIA στην Πολωνία. Έχει γραφτεί το άρθρο αυτό από δύο δημοσιογράφους οι οποίοι έχω εμπλακεί εδώ και χρόνια στην περίπτωση, τον κύριο Άνταμ και τον Βόιτσα Ζουκνόφσκι οι οποίοι λέγουν ότι υπήρξαν επίσημες κατηγορίες προς τον κύριο Σεμανκόφσκι ο οποίος στην εποχή των ε, φυλακών της ε, CIA ε, ήταν ο υπεύθυνο των μυστικών υπηρεσιών στην Πολωνία. Οι κατηγορίες αυτές έχουν υποβληθεί εναντίον του από τον Ιανουάριο του 2012. Σύμφωνα όμως με την πολωνική νομοθεσία υπάρχει μία διαδικασία που επιτρέπει προφορικές επερωτήσεις βάσει εγγράφων που έχουν προϋποβληθεί και οπότε ο ο ενδιαφερόμενος μπορεί ε, να παρουσιάσει στοιχεία βάσει των κατηγοριών και ο κύριος Σιμαρκόνσκι ε, ζήτησε να του ε, χορηγηθεί αυτό το καθεστώς και εντωμεταξύ η έρευνα έχει μετατεθεί από το εφετείο της βασοβίας στο εφετείο της Κρακοβίας. Νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο βασικά στοιχεία τα οποία έχουμε στη συνέχεια αυτού του άρθρου το οποίο επίσης μας, μας προδιαθέτει ότι υπήρξε έφεραν και άλλες υπηρεσίες στην Πολωνία που έχουν εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά σαν ε, νομικό σύμβουλος μη κυβερνητικών οργανώσεων ε, ε, η δυνατότητά μου κινήσεων είναι περιορισμένη και μπορώ εδώ απλούστατα να αναφερθώ εις τις κατηγορίες που έχουν δημοσιευτεί επίσημα στον πολωνικό τύπο. Ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Τώρα έχουμε την ε, τρία, τρίτη παρουσίαση της κυρίας Άμπριτ Σίνγκ, ε, κυρία νομομαθή Εθνικής Ασφαλείας και Αντιτρομοκρατικής Δράσης της ε, Open Society Justice Initiative σχετικά με τις περιπτώσεις Ελ Μασρί και Αλ Νασρίμπη θυμάτων έκδοσης και, της, και μυστικής κράτησης στην Ευρώπη. Ευχαριστώ, χαίρομαι που είμαι εδώ. Είμαι νομομαθής στο, Open Society Justice Initiative, που είναι μια οργάνωση που εκπροσωπεί τον Ελ Μάστρι, που είναι Γερμανός ε, υπήκος, ε, και τον ε, Αλ Νασίρι, που είναι Σαουδάραβας. Έχουν υποβάλει και δύο αμηνήσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η υπόθεση του Γερμανού υπηκόου Ελ Καλέντ Ελ Μασρή δείχνει την συνοχή της Μακεδονίας ε, και στην υπόθεση του Σαουδάραβα Αμπν Αλ Νασίρη δείχνει την ε, ε, συνοχή της Πολωνίας σε αυτό το πρόγραμμα. Και πρόσφατα ε, μαθεύτηκε ότι και η Ρουμανία συνεργάστηκε για την κράτηση του Αλ Νασίρη. Τώρα έχουμε κάποια στοιχεία για την υπόθεση Έλμα Μασρή. Τον, 31 Δεκεμβρίου του 2003 ο κύριος Έλμα Μασρή ε, ταξίδευε από τη Γερμανία στα Σκόπια με Πούλμαν ε, και έφτασε στα σύνορα. Όταν έφτασε στα σύνορα, ε, αξιωματούχοι των διοκτικών αρχών της Μακεδονίας κατάσχεσαν το διαβατήριό του και τον κράτησαν για πολλές ώρες. Η συνεχεία μεταφέρθηκε από ένοπλους ε, σε πολιτικά ε, στο Σκόπι ε, μερά ξενοδοχείο στα Σκόπια, όπου κρατήθηκε, χωρίς να ξέρει κανένας που βρίσκεται, από τις μακεδονικές αρχές για 23 μέρες, τον ε, φύλαζαν 24 ε, ώρες 24 ώρο ένοπλοι αξιωματικοί Μακεδόνες σε βάρδιες. Οι κουρτίνες ήταν κλειστές μέρα και νύχτα και δεν μπορούσαν να φύγει από το δωμάτιο. Τον ανέκριναν κατ' επανάληψη και του είπαν να παραδεχτεί ότι ήταν μέλος της Αλκάιντα. Ε, ζήτησε κατ' επανάληψη να δει ένα δικηγόρο, έναν μεταφραστή, έναν υπάλληλο του γερμανικού προξενείου, να έρθει σε επαφή με την οικογένειά του, με την γυναίκα του, αλλά του είπαν όχι. Και μια φορά που πήγε προς την πόρτα και προσπάθησε να φύγει, τρεις από τους δεσμοφύλακές του ε, τον σημάδεψαν με ένα όπλο και απείλησαν να το σκοτώσουν. Ε, στις 23 Ιανουαρίου 2004, 7 ή 8 Μακεδόνες Μπήκαν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, το, του βάλαν ε, χειροπέδες, του δίσαν τα μάτια, τον έβαλαν σε ένα αυτοκίνητο και τον πήγαν στο αεροπλάνο, στο αεροδρόμιο του, των Σκοπίων. Ε, τον έβγαλαν από το αυτοκίνητο, πάντα με τις χειροπέδες, ε, τον έβαλαν σε ένα κτίριο ε, όπου το κακομεταχειρίστηκαν και εν συνεχεία τον ανάγκασαν να μπει σε ένα αεροπλάνο της CIA και πήγε με το αεροπλάνο στο Αφγανιστάν. Εκεί τον κράτησαν για τέσσερις μήνες και υπέστη βασανιστήρια σε ένα, σε ένα κέντρο κράτηση της CIA που είναι γνωστό Salt Pit. Ε, μέχρι τις 28 Μαΐου 2004 εκεί Εν συνεχεία τον άφησαν ελεύθερο κάπου σε ένα ηρεμικό μέρο ε, και απόμερο μέρο στην Αλβανία χωρί καμία εξήγηση. Αυτό που είναι ενδιαφέρον για αυτή την υπόθεση είναι ότι είναι προφανέ ότι ο κύριο Αλμασρή είναι προφανώ ε, αθώο. Η γερμανική κυβέρνηση μάλιστα ε, παραδέχτηκε ότι ήταν αθώος. Στις 6 Δεκεμβρίου του 2005 η γερμανική καγκελάρ, καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ δημοσία δήλωσε μετά από συνάντηση που είχε με την Αμερικανίδα Υπουργό Εξωτερικών Κοντολίζα Ράι ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, παραδέχτηκαν ότι είχαν κάνει λάθο την υπόθεση του Ελ Μάστρι. Μετά από ε, επίσημε έρευνε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από το Συμβούλιο τη Ευρώπη και από την Bundestag, επιβεβαιώθηκε ε, ακριβώ αυτή η ιστορία του κύριου Ελ Μάστρι. Παρά το γεγονό αυτό, τα 8 χρόνια που μεσολάβησαν, από την δοκιμασία του κύριου Ελμάστρη, σε αυτά τα 8 χρόνια ούτε οι Αμερικανοί ούτε η μακεδονική κυβέρνηση παραδέχτηκαν το ρόλο τους στην διαδικασία αυτή έκδοσης, απαγωγής κτλ. Ούτε ζήτησαν συγγνώμη, ούτε του έδωσαν αποζημίωση. Η μήνυση που έκανε αντίον των Ηνωμένων Πολιτειών ε, δεν έγινε παραδεκτή γιατί ήταν υποτίθεται κρατικό μυστικό και η κυβέρνηση της Μακεδονίας αρνήθηκε την εμπλοκή της στην υπόθεση. Ε, ούτε επίσης ε, η μακεδονική κυβέρνηση έκανε αποτελεσματική έρευνα για να διερευνήσει τους ισχυρισμούς του Ελ Μάστρι. Στις 6 Οκτωβρίου 2008 ο Ελ Μάστρι υπέβαλε επίσημο αίτημα στο γραφείο του εισαγγελία των Σκοπίων για να διεργηθεί ποινική έρευνα εναντίον της παράνομης κράτησης και της απαγωγής και να ξεκινήσει ποινική διαδικασία εναντίον των υπευθύνων. Ε, όμως ε, δεν έγινε τίποτα από την κυβέρνηση της Μακεδονίας και πέρασε το χρονικό όριο παραγραφής αρχές του 2009. Τον Ιανουάριο του 2009 ε, υποβλήθηκε παρόμοια αστική αυτή τη φορά μήνυση για αποζημίωση ε, εναντίον του Μακεδονικού Υπουργείου Εσωτερικών λόγω της παράνομης απαγωγής ε, η υπόθεσή του ακόμα εκκρεμεί, δεν έχει γίνει τίποτα. Και ούτω ή άλλω με αυτή την αστική διαδικασία δεν μπορεί να υπάρξει ε, επανόρθωση για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων. Το, η, το Σεπτέμβριο του 2009 η οργάνωσή μου ε, υπέβαλε μία μήνυση ε, κατά της Μακεδονίας στο, ανθρώπινο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, γιατί θεωρείται ότι η Μακεδονία έπαιξε το ρόλο της αυτή την, στα βασανιστήρια, στην παράνομη κράτηση και έκδοση του Ελμάστρη. Ε, στο αίτημα αυτό που έχει υποβληθεί, ο Ελμάστρη προσπαθεί να πετύχει την αποκατάσταση της αλήθειας. Ε, η αίτηση αυτή διαβιβάστηκε στη μακεδονική κυβέρνηση τον Οκτώβριο του 2010 και τον Ιανουάριο του 2012, ε, κατά την αγνώριση της σημασίας του, της υπόθεσης, η υπόθεση αυτή πήγε στο σώμα Μίζωνος συνθέσεως ε, που θα συνεδριάσει στις 16 Μαΐου του 2012. Η δεύτερη υπόθεση που θα ήθελα να σας περιγράψω είναι η περίπτωση του Αμπ Αλ Ραχίμ Αλ Νασίρι, και γίνεται λόγος για τη συνενοχή της ε, πολωνικής και ρουμανικής ε, κυβέρνησης ε, στο αυτό το πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αλνασίρη εχμαλωτίστηκε και μεταφέρθηκε σε φυλακή της CIA ε, μεταφέρθηκε στο Αφγανιστάν, στο Σολτ Πιτ και τον κράτησαν επίσης και στην ε, Μπανκόκ, σε μυστική φυλακή στην Ταϊλάνδη, ε, όπου εκεί τον ανέκριναν πολύ βία. Ξέρετε, με αυτό το βασανιστήριο του εικονικού πνιγμού, Εν συνεχεία, στις 5 Δεκεμβρίου του 2002 η CIA μετέφερε τον κύριο Αλνασίρη στην μυστική φυλακή στην Πολωνία με τη βοήθεια των πολωνικών αρχών που προσέφεραν εντυπωσιακά επίπεδα ασφάλειας ε, για τις πτήσεις που έκαναν αυτή τη μεταφορά του. Στην Πολωνία, Αμερικανοί ανακριτές ε, υπέβαλαν τον Έλληνα Σύρη σε εικονική εκτέλεση ε, με ηλεκτρονικό τρυπάνι. Αυτός ήταν γυμνός και κουκουλωμένος κοπανούσαν ένα αυτόματο όπλο κοντά στο κεφάλι του, ο ίδιος ήταν αλυσοδεμένος μπροστά τους και απειλούσαν ότι θα φέρουν τη μητέρα του για να την βιάσουν μπροστά του. Αυτά βρίσκονται σε επίσημα έγγραφα των Αμερικανών και περιγράφουν ακριβώς αυτά τα γεγονότα. Κατά τη διάρκεια αυτής της ε, χρονικής περίοδου που ήταν κρατούμενο στην Πολωνία. Στι 6 Ιουνίου 2003 η Πολωνία βοήθησε τι ΗΠΑ ούτω ώστε να μεταφέρουν μυστικά με αεροπλάνο ε, τον Αλνασίρι εκτό Πολωνίας παρά το σοβαρό κίνδυνο να υποστεί και άλλα βασανιστήρια, να κρατηθεί χωρί να ξέρει κανένα που είναι, ε, να υποστεί άδικη δίκη και να αντιμετωπίσει και το ενδεχόμενο της θανατικής ποινής ε, στην Αμερική. Αυτό που είναι σημαντικό με αυτή την υπόθεση είναι ότι φυσικά Ξέρουμε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ σχεδόν παραδέχτηκε ότι κράτησε μυστικά διάφορους φυλακισμένους ε, στο εξωτερικό και ε, παραδέχτηκε ότι χρησιμοποίησε σκληρές τεχνικές ανάκρισης και βασανιστήρια. Ε, δέχτηκε ότι χρησιμοποίησε αυτή, αυτό το βασανιστήριο του εικονικού πνιγμού σε τρεις ε, φυλακισμένους. ο κύριος Μπλακ προηγουμένως είπε προηγουμένως ότι Αυτές ε, οι πληροφορίες είναι γνωστές, τις έχουν ε, παραδεχτεί οι Αμερικανοί. Νομίζω ότι είναι και η ώρα πια να αναγνωριστεί ότι κάποια πράγματα δεν αμφισβητούνται πια. Είναι αδιαμφισβήτητα γεγονότα και στοιχεία. Και το πρόγραμμα μυστικών κρατήσεων είναι ένα από αυτά τα στοιχεία. Το, δέχτηκε, το παραδέχτηκε στις, ε, το Σεπτέμβριο, στις 6 του Σεπτεμβρίου του 2006 ο πρόεδρος Μπούς. Κάποια στιγμή μεταξύ του 2003 και του 2006 ο κύριος Αλνάσρη ε, υπέστη μυστική κράτηση σε μια άλλη ε, φυλακή μυστική στη Ρουμανία. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί σε μια δήλωση του Ιουνίου του 2011 σε έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ε, υπάρχουν και άλλες ε, πηγές που το πιστοποιούν. Η Τζούλια Χολ το ανέφερε στην παρουσίασή της. Και στην γερμανική κυβέρνηση επίσης, σε μια εκπομπή, επιβεβαιώνεται η ακριβής τοποθεσία της φυλακής όπου κρατήθηκε ο κρατούμενος αυτός. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω λίγο πίσω και να σας πω ότι αυτή η υπόθεση είναι σημαντική όχι μόνο γιατί αφορά μια παράνομη κράτηση ενός ανθρώπου που κανένας δεν ήξερε που είναι, όχι μόνο γιατί ε, ο άνθρωπος αυτός ε, υπέστη βασανιστήρια σε ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά και γιατί σχετίζεται και με την υποχρέωση, όπως λέει το Συμβούλιο της Ευρώπης, να μην ε, επιτραπεί η μεταφορά φυλακισμένων, ε, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να βασανιστούν εκεί που θα πάνε και να ε, υποστούν την εσχάτη των ποινών. Και η υπόθεση του ανθρώπου αυτού είναι η πρώτη υπόθεση θαντικής ποινής που θα εκδικάσει στατιωτικό δικαστήριο, στατιωτική επιτροπή ουσιαστικά στο Γκουαντάναμο, που δεν είναι ανεξάρτητο δικαστήριο και έχει κανόνες λειτουργίας που διαφέρουν πάρα πολύ από αυτές των νομοσπονδιακών δικαστηρίων και που επιτρέπει ε, να κατατεθούν στοιχεία τα οποία τα έχουν ε, αποσπάσει με πολύ σκληρές μεθόδους Κάτι που ήταν πρακτική σε αυτό το πρόγραμμα. Επίσης, ε, κάποια πρακτικά, ε, τα οποία όμως τα έχουν χτενίσει πάρα πολύ ε, το 2007, που πήραν από από ανάκριση στον Κουαντάναμο αποκαλύπτουν ότι ο Αλνασίρη είπε ότι τα πέντε χρόνια που κρατούμε με βασανίζουν. τη μία φορά με βασανίζουν με τον έναν τρόπο, την άλλη φορά με έναν άλλο τρόπο. Ε, με βάση την περιγραφή του Αλνασίρη για τα βασανιστήρια, ε, ο ίδιος δηλώνει ότι υποθύμησε από τα βασανιστήρια. Είπε ότι πριν ε, με συλλάβουν ε, μπορούσα να τρέχω 10 χιλιόμετρα. Τώρα δεν μπορώ να περπατήσω πάνω από 10 λεπτά. Τα νεύρα μου είναι πρισμένα μέσα στο σώμα μου. Αυτό είναι το μόνο ε, στοιχείο το οποίο δήλωσε ο ίδιος και το οποίο έχουμε στα χέρια μας. Ε, ε, το άλλο γελίο στοιχείο αυτής της υπόθεσης είναι, όπως είπε και ένας Αμερικανός δικηγόρος, ότι όλες αυτές οι υποθέσεις είναι διαβαθμισμένε και οτιδήποτε πει είναι διαβαθμισμένο και δεν μπορεί κανένα ούτε μέσω των δικηγόρων του να απευθυνθεί στο, στον κόσμο, να μιλήσει για τα φρικόδη βασανίστρια τα οποία υπέστη. Υπάρχουν πολλαπλά στρώματα ε, παραβιάσεων. Έχετε βασανιστήριο, ε, σκάτη των ποινών, ε, άδικη δίκη από μη ανεξάρτητο δικαστήριο και επίσης έχετε και την ομερτά, έχετε τη φήμωση του, φυλακισμένου, ο οποίος δεν μπορεί καθόλου να μιλήσει για το τι του συνέβη. Στις 20 Απριλίου του 2011 η Στρατιωτική Επιτροπή και οι εισαγγελεί τη ε, απήγγειλαν κατηγορίε εναντίον του Σύρι ε, για τον υποτιθέμενο ρόλο του στην ε, επίθεση του USS Cole το 2000 και για την επίθεση του γαλλικού δεξαμενόπλου, αστικού δεξαμενόπλου, MV Limburn, στον κόλπο του Άντεν το 2002. Η... Η στρατιωτική αυτή επιτροπή δέχτηκε αυτές τις κατηγορίες και τώρα αντιμετωπίζει την εσχάτη των ποινών ο φυλακισμένος. Δεν υπάρχει περίπτωση να υποστεί δίκαιη δίκη, αλλά μπορεί να, μετά τη δίκη αυτή να καταδικαστεί σε θάνατο. Ε, η πολωνική και η ρουμανική κυβέρνηση ε, είναι συνυπεύθυνε γιατί επέτρεψαν τη μεταφορά τους παρά το γεγονός ότι υπήρχε ο κίνδυνος για την ασχάτη των ποινών. Μία πολωνική ε, ποινική διαδικασία ξεκίνησε εδώ πέντε χρόνια μετά της, ε, τη συλλογή αδειάστων στοιχείων για το ρόλο της Πολωνίας και ε, εδώ και τέσσερα χρόνια ε, δεν υπάρχει πρόοδος. Δεν είναι διαφανής αυτή η έρευνα και σε ό,τι αφορά τον πελάτη μου δεν υπάρχει σημάδι προόδου, δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθεί, υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητά της. Το Μάιο του 2011 η Open Society Justice Initiative υπέβαλε μία αίτηση ε, εκ μέρους του Al-Nashri στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, για την συνοχή της Πολωνίας ε, στην κράτησή του, χωρίς να ξέρει κανένας που είναι, και τη μεταφορά από την Πολωνία παρά τους σοβαρούς κινδύνους για βασανιστήρια, κακομεταχείριση και θανατική ποινή. Οι αιτήσει αυτέ ε, ζητούν από την πολωνική κυβέρνηση να χρησιμοποιήσουν πάρα αυτά όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους ε, για να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υποστεί την εσχάτη των πίνων ο Αλνασίρη ε, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διπλωματικές διαβεβαιώσεις από τις ΗΠΑ ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Τι σημαίνουν όλα αυτά για το, αυτές οι δύο υποθέσεις μάλλον για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με βάση τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της α, ε, ανθρώπινης ζωής, του, ε, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου κτλ. Η συμπεριφορά της Μακεδονίας ε, στην περίπτωση του Ελνασίρη ε, παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και θέτει ερωτήματα για την καταλληλότητα της Μακεδονίας για προσχώρησή της στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να διερευνήσετε ακριβώς αυτή την υπόθεση. Πολωνία και Ρουμανία τώρα. Ε, είχαν στο ταφό τους τέτοιες μυστικές φυλακές και επομένως ε, αψηφούν τις αρχές που υπάρχουν στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να διενεργήσουν αποτελεσματικές έρευνες και να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή του, ούτω ώστε να εξασφαλίσουν ότι ο Ελνάσουρι δεν θα υποστεί την ασχάτη των ποινών. Το πιο σημαντικό είναι, αυτά είναι δύο απλώς παραδείγματα ανθρώπων των οποίων τα δικαιώματα έχουν παραβιαστεί ε, σε, αυτό σε, αυτή, την σε αυτή την συνενοχή με τους Αμερικανούς. Ε, στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αφορούσε πολύ περισσότερα άτομα και όπου συστηματικά γινόταν παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τώρα την ευκαιρία να παίξει τον ηγετικό ρόλο, ούτω ώστε να υπάρξει λογοδοσία για τι εκδόσει αυτέ. Ε, για να δείξει στι ΗΠΑ ότι η Ευρώπη είναι διαφορετική. Ότι οι ΗΠΑ μπορεί να μην θέλουν να κοιτάξουν πίσω και να δουν τι έκαναν ακριβώ με τα βασανιστήρια, αλλά ότι η Ευρώπη είναι πιο ανθεκτική από αυτό και δεδομένων των πολλών ευρωπαϊκών χωρών που ήταν ε, συνένοχοι με τους Αμερικανούς, ε, νομίζω ότι η Ευρώπη τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι, ούτως ώστε να μην πάρουν οι Αμερικανοί μέσα από τη μάζα των κρατών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποιες χώρες ε, και τις, τις απομονώσουν και τις ε, τιμωρήσουν γι' αυτό, ούτω ώστε να πριτανεύσουν οι αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις ομιλητές. Τώρα έχουμε κι άλλο κατάλογο με ομιλητές. Προτείνω να κάνουμε το εξής. Σας είπα ότι κάποιοι από τους εθνικούς φορείς που είχαν προσκληθεί εδώ δεν ε, μπόρεσαν να έρθουν. Όμως, πολύ σύντομα θα σας πω τι μας έχουν στείλει και μετά θα περάσουμε στον δεύτερο γύρο παρουσιάσεων και να μην ξεχνάμε παρακαλώ ότι στις 12 πρέπει να ψηφίσουμε. Οπότε ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε ολοκληρώσει στις 12. Όπως ε, σας έλεγα και πριν έχουμε πέντε ομιλητές με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή από τη Δανία, την Πολωνία, τη Λιθουανία, τη Ρουμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο σε δικαστικό επίπεδο και θα συνοψίσουμε τι μας είπανε. Ο κύριος Αντρέ Σέρεμετ, που είναι Γενικός Αγγελέας της ε, Πολωνίας, μας λέει ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εξηγεί τους λόγους που δεν μπορεί να είναι εδώ μαζί μας σήμερα και λέει ότι τα στοιχεία που έχουν ε, μαζευτεί από το 2008 από τους ε, συμμετέχοντες στην έρευνα για τις παράνομες αυτές κρατήσεις κτλ. είναι απόρριτες. Τα περισσότερα στοιχεία λοιπόν είναι απόρριτα. Τι ακριβώς λέει. Λέει ότι τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις μαρτυρίες των μαρτύρων είναι ε, κρίνονται top secret, απόρριτα. Και συνεπώς που σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και να συζητηθούν εδώ και ότι όποιος ε, χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία και τα παρουσιάσει είναι ένοχος. Τέτοιου λοιπόν διαβαθμισμένες πληροφορίες δεν πρέπει να κυκλοφορούν και έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό η συγγελία. Στις περισσότερες σοβαρές περιπτώσεις υπάρχουν ε, ε, βέβαια δικαστικές διαδικασίες στην Κρακοβία και ό,τι μέτρο ε, λαμβάνεται ε, για να μην είναι απόρριτες αυτές οι πληροφορίες εφόσον προχωρήσει αυτή τη διαδικασία και δεν είναι διαβαθμισμένε οι πληροφορίε αυτέ θα ενημερωθούμε. Ο κύριο Τόμα Βίκλερ τώρα, ο οποίο είναι ο νομικός σύμβουλος της νομικές υπηρεσίε της Δανίας, του Υπουργείου Εξωτερικών, είναι πρέσβή στην Αμερική και λέει ότι θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε εφόσον είναι δημόσιος υπάλληλο να συμμετέχει σε μια τέτοια συνάντηση σαν τη σημερινή, εφόσον το Ινστιτούτο της Δανίας εκπονεί έκθεση αυτήν την εποχή όσον αφορά τις, τους ισχυρισμούς για μυστικές φυλακές κλπ. Ο κύριος Τότορ Μιλανέσκου από την Ρουμανική Γερουσία έχει επίσης προσκληθεί εδώ ως πρόεδρος της Επιτροπής για τη Δημόσια Ασφάλεια της Ρουμανικής Γερουσίας, μας λέει, θέλω να ενημερώσω την Επιτροπή σας, Λίμπε, ότι η εντολή μου λύγει. Και ο επόμενος πρόεδρος, ο κύριος Μπόκερ Κολέ, δυστυχώς δεν μπορεί να παρευρεθεί στην ακρόαση αυτή. Ο Σερ Πίτερ Κίψον τώρα από την Ερευνητική Επιτροπή του Ηνωμένου Βασιλείου ε, μας ενημερώνει ότι λυπάται που δεν μπορεί να είναι εδώ αλλά λέει ότι τον Ιανουάριο θα υπάρξουν συμπεράσματα όσον αφορά την περίπτωση δύο Λίβιων και για τις μυστικές κρατήσεις και βασανισμούς που υπέστησαν. Ο κύριος Ελβάσκας τώρα, που είναι πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Λιθωνίας, αρμόδιος για τα θέματα αυτά, επίσης μας λέει ότι έχουν ότι έχει υπάρξει έρευνα και βάσει των στοιχείων που έχει τώρα η Επιτροπή μέχρι τώρα δεν υπήρξαν κρατήσεις ή βασανισμοί στο εικαζόμενο αυτό μέρος. Όσο τη μεταφορά ε, επίσης από τη CIA κρατούμενων η Επιτροπή δεν έχει καταλήξει σε τέτοιο συμπέρασμα. Υπάρχουν διάφορα έγγραφα στη διάθεσή σας. Χωρίς άλλη καθυστέρηση λοιπόν και άλλα σχόλια, τώρα θα συζητήσουμε. Κυρία Μπέγαρα, είναι η πρώτη που έχει στήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ που οργανώσατε την ε, συνάντηση αυτή. Έχω να κάνω δύο σύντομα σχόλια. Πρώτα απ' όλα, Σας άκουσα να περιγράφετε την πραγματικότητα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίσετε στην έρευνά σας. Και μετά άκουσα αυτά που είπατε εσείς, Πρόεδρε, γιατί δηλαδή οι διάφοροι εθνικοί φορείς σχετικοί με τις έρευνες αυτές δεν μπόρεσαν να έρθουν. Ε, νομίζω ότι όλα όσα γίνονται για αυτή την υπόθεση ξεπερνούν τον Κάφκα κατά πολύ. Είναι σαν να πρόκειται για άλλο κόσμο. Έχω όμως να πω και κάτι για την χώρα μου, την Ρουμανία, όπου οι ισχυρισμοί τέτοιοι υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό. Όμως δυστυχώς δεν υπάρχει πραγματική έρευνα που να λαμβάνει η χώρα. Έγινε κάποια έρευνα από το Κοινοβούλιο κάποια στιγμή που εξέφρασε τις περιορισμένες τις δυνατότητες, αλλά Κατά τη γνώμη μου, αυτό που φταίει είναι η άρνηση της κυβέρνησης και των ε, αξιωματούχων. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πρόκειται δηλαδή για αδιαφορία. Η αλήθεια είναι ότι στην χώρα μου, αντίθετα από ό,τι συμβαίνει με την Πολωνία, δεν υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες να ασχολούνται με αυτό το θέμα, ούτε και δημοσιογράφοι οι οποίοι να προσπαθούν να καταλήξουν σε, κάποια, σε κάποιο συμπέρασμα στην Πολωνία, αν μη τι άλλο έχει ξεκινήσει μία εισαγγελική έρευνα. Σε μας όχι. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι έρευνας εκτός από το κοινοβουλευτικό. Έχω όμως και μία ερώτηση, παρακαλώ και λυπάμαι που δεν είναι εδώ ο κύριος Γιώτης. Ήθελα κάτι να τον ρωτήσω. Θα ρωτήσω λοιπόν ανταυτού τον κυρί... την κυρία Σίνγκ. Δεν λέω ότι θέλω να μου αποκαλύψετε τις πηγές της έρευνά σας, αλλά η ερώτησή μου έχει να κάνει με το κτίριο που φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε για τις ανακρίσεις έχετε πηγές μέσα από τη χώρα ή εκτός της χώρας. Αυτή είναι η μόνη ερώτηση στην οποία θέλω να μου απαντήσετε. Ευχαριστούμε. Κύριε Κοαγιό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αλλά η ομάδα η οποία είχε καταρτιστεί ήταν ε, πολύ ε, ε, αλληλεγγύη και ο εισηγητής Φκλάντιο Φάβα, η Σεσίλια Μάλστρεμ και τα υπόλοιπα μέλη είχαν πολύ καλή συνεργασία μεταξύ τους αλλά είχαμε αντιληφθεί ότι υπάρχει, υπήρχε αποσιώπηση ορισμένων ε, γεγονότων και δεν με εκπλήσει ε, αυτά τα οποία λέγονται ιδίω για την Πολωνία διότι η αντιπροσωπεία μας είχε μεταβεί στην Πολωνία και είδαμε ότι είναι μία χώρα όπου όλες οι αρχές αρνήθηκαν να μας ε, αντιμετωπίσουν. Η μόνη χώρα όπου πήγαμε και μας συμπεριφέρθηκαν έτσι ήταν η Πολωνία. Ε, πήγαμε και στη Washington, στις Αμερικανικές αρχές και σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει αυτή η τρομερή σιωπή και διαιωνίζεται η κατάσταση. Σχετικά με το Ευρωκοινοβούλιο, χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα και χαίρομαι που γίνεται αυτή η ακρόαση, αλλά το πρώτο εγγραφό το οποίο υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν το Σεπτέμβριο του 2007, οπότε αποφασίσαμε ότι θα υπήρξε και ανακίνηση του θέματος και είχα στείλει μία επιστολή στον πρόεδρο Λόπες Αγγιλάρ ε, από το 2010 και τώρα ξεκινάει η διαδικασία αυτή διότι υπήρξαν ορισμένα προβλήματα σχετικά με την διεκπαιρέωση ε, της υποθέσεως αυτής υπήρχε ε, ένας φαύλος κύκλος που μας εμπόδιζε να προχωρήσουμε και τώρα βλέπουμε τα άτομα τα οποία έχουν εξαιρετική επίδοση στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωνάτων και μπορούν να μας βοηθήσουν αλλά θα ήθελα να περιοριστούμε ε, σε ε, αποδεδειγμένα περιστατικά για να είμαστε αξιόπιστοι. Διότι όταν ξεκινήσαμε πολλοί μας είπαν ότι όλα αυτά ήταν ψεύτικα και ε, ό,τι λέγαμε για έκτακτες παραδόσεις στη CIA ήταν ψευδή. Αλλά από το 2006 ο Τζόρτζο Μπούς παραδέχτηκε αυτές τις κινήσεις και του ε, ε, βασανισμούς. Όλα δηλαδή τα οποία είχαμε πει εδώ και που πολλοί ε, μας κατηγορούσαν ότι ψευδόμεθα έχουν αναγνωριστεί από τον George Bush. Ξέρουμε ότι αυτά συνέβησαν και ότι υπάρχουν ορισμένοι που απορρίπτουν την ύπαρξη βασανισμών αλλά θέλω να πω στην κυρία Φλότρο ότι παρόλο που είναι βασικό να συγκεντρώσουμε στοιχεία πρέπει να κάνουμε τα σωστά ερωτήματα προς τα κράτη-μέλη και να δούμε κατά πόσο εφήρμοσαν τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί εμείς είχαμε διατυπώσει ε, ε, συστάσεις για τη σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείες, για την αντιμετώπιση των μυστικών υπηρεσιών, για την παρακολούθηση των αεροπορικών πτήσεων για την εφαρμογή των ψηφισμάτων μας και υπάρχει και, ε, το, και η σύμβαση του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια. Όλα αυτά τα οποία εμείς θεωρούσαμε βασανιστήρια θεωρούνται από την ε, κυβέρνηση Μπούς ότι δεν ήταν βασανιστήρια κατά κάποιο περίεργο τρόπο. Δεδομένου λοιπόν των σχέσεών μας με τις χώρες αυτές θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θέσει τα ερωτήματα προς τα κράτη-μέλη και να τους ρωτήσει εσείς τι έχετε κάνει για να εφαρμόσετε αυτές τις συστάσεις και αν δεν έχει γίνει τίποτα θα είναι σκόπιμο αυτό να τοποθετηθεί στην ε, έκθεσή μας. Σας ευχαριστώ κύριε Κοέγιο. Ο χρόνος είναι περιορισμένος και θα έπρεπε σε δύο-τρία λεπτά να έχει περιοριστεί ο καθένας διότι έχουμε ψηφοφορία στις 12 και είναι ε, κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν ε, καταλαβαίνουν τι συμμετέχοντες στην Επιτροπή Ελευθεριών. Οι συμμετέχοντες στις ψηφοφορίες έρχονται ακριβώς την ώρα που πρέπει με την κάρτα τους για να ψηφίσουν και εκνευρίζονται αν δεν μπορούν να οργανωθούν οι ψηφοφορίες εν γέρος. Έχουμε ακόμη και τις ερωτήσεις και τα σχόλια της κυρίας Φλότορ και του, της κυρίας Λατφόρντ, η κυρία Γκόμες τώρα. Ευχαριστώ. Τηλεγραφικά, ο τίτλος της έκθεσης θα πρέπει να είναι «Μυστικές και παράνομες αμερικανικές κρατήσεις, πρόγραμμα αμερικανικών κρατήσεων ε, στην Ευρώπη». Δεν είναι μόνο η CIA, είναι στρατιωτικό πρόγραμμα, δεν είναι μόνο αεροπλάνα, είναι και πλοία ε, και πρόκειται για κέντρα κράτησης. Έχει όλα αυτά τα στοιχεία αυτό το πρόγραμμα. Και φυσικά ε, έχει και βασανιστήρια. Έχουμε θύματα. Προηγουμένως ε, κάποιος ρώτησε ε, τι στοιχεία έχουμε. Έχουμε θύματα. Θύματα, ο ε, όπως ο Αμπού Ζουμπάιντα, που είναι ακόμα κρατούμενοι και άλλοι που είναι ακόμα, βασανίζονται ακόμα από αυτά που υπέστησαν. Ο κύριος Κοέλιο είπε ότι το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο. Γι' αυτό υπήρχε όλη αυτή η αντίδραση. Ορισμένοι προασπίστηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Και η συνενοχή φτάνει ως την κορυφή. υπάρχουν υψηλότερες πολιτικές ευθύνες ως το υψηλότερο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Θα γίνει μια αποστολή στη Λιθουανία σύντομα. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσθέσουμε και την Πολωνία με βάση τα στοιχεία που έχουμε. Και κάποια στιγμή και να πάμε και στη Ρουμανία. Θα είναι πολύ σημαντικό, εστιάζουμε σε κάποιες χώρες για τις οποίες έχουμε περισσότερα στοιχεία ε, γιατί η αποκάλυψη αυτών των υποθέσεων ε, θα έχει επιπτώσεις και για άλλες χώρες επίσης, οι οποίες επίσης θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Άλλες, άλλα κράτη-μέλη δηλαδή. Ε, είναι σημαντικό ότι να ζητήσουμε να δούμε και τους πολιτικούς, τους υπεύθυνου υπουργού και τους υπεύθυνου των μυστικών υπηρεσιών. Μια φορά στην Πορτογαλία η Επιτροπή μας ζήτησε να δει τον Υπουργό Άμυνας που είναι τώρα Υπουργό ε, Οικονομικών τη Πορτογαλία. Αρνήθηκε να μιλήσει στην κοινοβουλευτική αποστολή όμω. Ζητήσαμε να μιλήσουμε με του επικεφαλεί των μυστικών υπηρεσιών και φυσικά ε, μα αρνήθηκαν την άδεια ε, να μιλήσουμε μαζί του. Αρνήθηκαν να μιλήσουν. Επίσης, το κόλπο να αλλάζει στον εισαγγελέα. Γίνεται μία έρευνα ε, και άλλα τον εισαγγελέα έθνη. Αυτό ε, ακριβώ έγινε και στην Πορτογαλία. Κλασικό κόλπο. Όταν μιλάω για την Πολωνία, δεν θέλω να μιλήσω χωρίς σεβασμό ε, για την χώρα αυτή. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σεβασμό προς τα, ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, δεν στρέφομαι εναντίον των Αμερικανών. με ενδιαφέρει αυτό το πρόγραμμα και που είναι εντελώς αντιαμερικανικό. Ευχαριστώ, κύριε Γκόμες. Κύριο Ποτρόφσκι. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση και είναι σημαντικό ότι η Επιτροπή μας, η Επιτροπή μας ασχολείται με αυτά τα θέματα. Εδώ μιλάμε όμως για κάποια ειδικά θέματα, για τις ε, υπηρεσίες πληροφοριών που υποτίθεται ότι προστατεύουν τα, τους στόχους των τρομοκρατών. Κυρία Σίγκα, που εσείς μιλήσατε για δύο υποθέσεις, του κυρίου Ελμάστρη, ας πούμε. Ο κύριος Ελμάστρη είναι ο ίδιος που ήταν εδώ ε, στο 2006 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με τον κύριο Κοέγιο εγώ μάλλον μαζί με τον κύριο Κοέλιο ήμουν τότε συντονιστή στην Επιτροπή. Ήταν ο ίδιος που είχε έρθει εδώ και μίλησε για αυτή την ιστορία. Μιλάμε για τον ίδιο. Ήταν φιλοξενούμενος μας το 2006 ο κύριος Ελμάστρη, αν δεν απατώμε. Το άτομο αυτό για το οποίο μιλάω εγώ ήταν Γερμανός υπήκος και επιβεβαίωσε ότι ανήκε σε μια οργάνωση που ε, βρίσκεται στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων και επιβεβαίωσε ότι έφερε όπλα και ότι η οργάνωσή του είχε όπλα. Είναι ο ίδιος Ελμάσρι, ο οποίος έφυγε από τη Γερμανία και πήγε στα Βαλκάνια. Και από ό,τι φαίνεται ισχυρίστηκε ότι πήγε ως τουρίστας ε, που η γυναίκα του επί έξι μήνες δεν ήξερε ότι εξαφανίστηκε. Ένας Γερμανός ε, που τον ανέκρινε μας είπε ότι απλώς ε, το θέμα αυτό ξεφούσκωσε. Είναι το ίδιο άτομο. Και θα ήθελα να σας πω το εξής. Α, ναι. Ε, δεν έχει νόημα να κοιτάμε μονομενες υποθέσεις. για μερικές υπάρχουν αμφιβολίες. Αυτός ο κύριος, ο κύριος Ελμάσουη, ήρθε εδώ το 2006. Έχει νόημα να αποκαλύπτουμε όλες τις λεπτομέρειες του αγώνα κατά της τρομοκρατίας, ένας αγώνας που σώζει ζωές. Έχει νόημα να προτάσουμε κάποιες αμφίβολες περιπτώσεις και την ίδια στιγμή να παραβιάζουμε τα δικαιώματα ανθρώπων που είναι οι στόχοι των τρομοκρατών. Και να μην ξεχνάτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε την έκθεση της Επιτροπής μας που λέει ότι δεν μπορεί να υποθεί πέραν πάση αμφιβολίας ότι στην Πολωνία υπήρχαν κέντρα κράτησης της CIA. Ευχαριστώ. Η σειρά σας κύριε Έντσιου. Το τελευταίο η τελευταία παρέμβαση πριν δώσουμε το λόγο και πάλι στους προσκεκλημένους μας. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Συμφωνώ με όλα όσα είπαμε εδώ. Έχω μια παρατήρηση και μια ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, στην Ρουμανία έχουμε κάνει πολλές έρευνες και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο αλλά και ανεξάρτητα μέσα. Και μετά από τις έρευνες αυτές δεν έχουμε καταλήξει σε συγκεκριμένο συμπέρασμα. Έχουμε μόνο εικασίες. Κυρία Σίνκ, πώς μπορείτε να είσαστε σίγουροι και να λέτε ότι στη Ρουμανία υπήρξε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι υπήρξαν παράνομα κέντρα βασανισμών. Τι αποδείξεις έχετε γι' αυτό. Μια στιγμή. Οι ομιλητές. Σύντομα. Να είσαστε σύντομοι γιατί αρχίζει να πιέζει ο χρόνος και πρέπει και να ψηφίσουμε στις 12. Συνεπώς, η κυρία Γιάκοψον πρώτα. Ή ο κύριος Μπότρου. Ο κύριος Μπότρου πρώτα, μάλιστα. Θέλω να... Θέλω να συμπληρώσω με ένα σημαντικό γεγονός, το οποίο είναι το εξής αυτό σχετικά με το σημερινό άρθρο στην Καζέτα Βαμπότσκα δηλαδή τη δυνατότητα να, υπάρξει μία αγωγή διότι η υπηρεσία των μυστικών υπηρεσιών έχει παραπέμψει τα θέματα του φακέλου των παρανών μετακινήσεων εις των Πολωνών Γενικό Εισαγγελέα παρόλο που δεν υπάρχει παραγραφή των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως ε, τα, η αποφυγή βασανιστήριων και ε, αν ε, συμβεί κάτι τέτοιο στην πολωνική επικράτεια θα έπρεπε το πολωνικό κράτος να έχει απαντήσει σε όλα αυτά και εντωμεταξύ υπάρχουν πάρα πολλές αποδείξεις ότι υπήρξαν φυλακές τη CIA στην ε, Πολωνία και ότι το θέμα εξετάζεται. Κυρία Σίνκ, θέλετε σύντομα να σχολιάσετε. Όσον αφορά την ερώτηση σχετικά με τον Χαλίντε Ελμάστρη που ήταν ε, ε, γερμανός υπήκος και είχε παρουσιαστεί εδώ, ίσως δεν καταλάβατε, δεν είχε κρατηθεί στη Ρουμανία ή στην Πολωνία, αλλά εις Τριφύρομ και αυτό σημαίνει ότι ε, οι ε, οργανώσεις πρέπει να παρακολουθούν τις υποθέσεις εάν εσείς είχατε κρατηθεί ε, σταλή σε μία παράνομη φυλακή στο Αφγανιστάν και είχατε βασανιστεί θα θέλατε το θέμα αυτό να παραπεμφθεί όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και από τους εισαγγελείς ε, ε, των εμπλεκομένων χωρών. Ο κύριος αυτός ε, δεν έχει αναλάβει καμία εγκληματική δράση. Η γερμανική κυβέρνηση παρεδέχθη ότι είχε κρατηθεί κατά λάθος πράγμα το οποίο ε, δηλώθηκε από τον Γερμανό υπεύθυνο μετά από συνάντηση με την Κοντολίζα Ράις. Και τέλος, όσον αφορά τις ε, έρευνες της ε, Ρουμανίας, λυπάμαι αλλά δεν ε, αρκούν ε, για να αντιμετωπίσουν ε, και να απαντήσουν στην μυστική κράτηση και τα βασανιστήρια και θέλω να σας αναφέρω ότι υπάρχουν οι εκθέσεις του Ντίκ Μάρτι το 2006 και το 2007 όπου λέγεται ευθαρσός ότι ε, υπήρξαν κέντρα στη Ρουμανία, ότι, ότι δημόσιες πηγές αποδεικνύουν ότι ο πελάτης μας κρατήθηκε στη Ρουμανία και όσον αφορά τις πηγές δεν μπορώ να σχολιάσω συγκεκριμένες εθνικές πηγές. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι υπήρχαν πολύ περισσότερες οι οποίες είχαν επιβεβαιώσει την ύπαρξη των φυλακών αυτών στην ε, ε, Ρουμανία. Η κυρία Λάτφορντ ως συντάκτρια της γνωμοδότησης ε, προς ε, την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για το θέμα αυτό το οποίο καλύπτει και η Επιτροπή Ελευθεριών. Δεν θέλω να σας παρεμποδίσω να ψηφίσετε. Θέλω να αποτύσω φόρο τιμή στους μη κυβερνητικού οργανισμούς και στους ε, δημοσιογράφους που ήταν πολύτιμοι τιμή βοηθή την τελευταία δεκαετία για να φτάσουμε στην αλήθεια. Και εγώ ενεπλάκη, ήμουν εισηγήτρια ε, για την έκθεση του Κοινοβουλίου για τον Κουαντάναμο ε, και το Σεπτέμβριο ε, του 2003 πήγα εκεί, ε, ήμουν αντιπρόεδρος της ε, προσωρινής επιτροπής, ε, ξέρω πολύ καλά τη δουλειά που έγινε. Ε, χαίρομαι που δουλεύω με την Ελέν Φλότ η οποία τώρα θα κάνει μια θαυμάσια δουλειά με την έκθεση αυτή. Το Υπουργείο Εξωτερικών ξέρω ότι σημείωσε ότι δεν απάντησε ε, στα αιτήματα αμοιβαία συνδρομής. Ε, την περασμένη εβδομάδα στη Ουάσιγκτον ε, συναντήθηκα με εκπρόσωπο του Υπουργείου ε, και του, τον ρώτησα γιατί συνέβη κάτι τέτοιο. Αυτά που ξέρουμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, απέτυχε πάταγωδός να εξασφαλίσει τη λογοδοσία από όλα όσα ξέρουμε που, ότι συνέβησαν. Ο Ζιλντε Κερκόφ την περασμένη εβδομάδα ε, προσυπέγραψε ένα άρθρο στο, στο European Voice και είπε τι όμορφη που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που τηρεί τα ανθρώπινα δικαιώματα στον, στην προσπάθεια καταπολέμησης της δημοκρατίας, εφαρμόζοντας την ποινική δικαιοσύνη. Είναι ηρωνία. Αν το δικαστήριο του Στρασβούργου, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σας παρακαλώ, γίνεται ακρόαση διακόπτη ο πρόεδρος. Εσείς στο βάθος, που είσαστε εντός της αίθουσας, τουλάχιστον να, να παραμείνετε σιωπηλοί, διότι κάποιος άνθρωπος μιλάει. Σας παρακαλώ, ήσυχα. Έλεγα λοιπόν, θα ήταν ηρωνία αν το δικαστήριο του Στρασβούργου ζητάει από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λογοδοτήσουν. Δεν περιμένω με ενπομονησία αυτές τις αποφάσεις, γιατί θα σηματοδοτήσω μία αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. το σχόλιο ότι πρέπει να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και να παραδεχτεί πράγματα που παραδέχεται η Αμερική είναι σωστό. Πρέπει να δούμε τι συνέβη και τι πρέπει να συμβεί στι Ηνωμένε Πολιτείες. Και το λέω αυτό και ως αντιπρόεδρος της ε, αντιπροσωπείας ε, σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Αμερικής. Κύριε Πεστρόφσκι, αν υπήρχαν, ε, αν υπήρχαν πραγματι... αν υπήρχαν ισχυρισμοί για τρομοκρατική δράση εναντίον του Ελ Μάσρι στην Ευρώπη, θα έπρεπε να υποστεί μια δίκαιη δίκη και όχι να κρατηθεί μυστικά σε φυλακές. Κυρία Φλότ, για να ολοκληρωθεί οι εργασία της ακρόασης. Ε, πολύ σύντομα, δεδομένε τη ώρα και τη κατάσταση, καταρχά θέλω να ευχαριστήσω όλου του παρεμβαίνοντε, γιατί νομίζω ότι σήμερα ε, βοήθησαν στον προβληματισμό μα, βοήθησαν στη σύνταξη τη θέση. Ε, δεν συζητάμε παλιέ ιστορίε ε, γραμμένες στα βιβλία της ιστορίας. Μιλάμε για μια επικαιρότητα καυτή, για γεγονότα επίκαιρα. Τρέχουν ακόμα οι έρευνε, τα θύματα δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμα. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε αποζημίωση για τις σοβαρότατες ε, πράξεις εναντίον τους. Από τις ομιλίες που ακούσαμε, η κατάσταση στην Πολωνία ε, τονίστηκε ιδιαίτερα. Ε, είναι και θέμα επικαιρότητα. Αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να ξεχνάμε την κατάσταση στις υπόλοιπες χώρες, Ρουμανία, Φερρυπίν. Για τη Ρουμανία ε, καλέσαμε έναν δημοσιογράφο ο οποίος ε, έγραψε ένα άρθρο ε, εντυπωσιακό για τις μυστικές φυλακές και τους χώρους μυστικών φυλακών στη Ρουμανία. Και παρότι η ρουμανική κοινωνία δεν είναι τόσο κινητοποιημένη, παρόλα αυτά υπάρχουν οι, οι οργανώσεις όπως η Χάπαντοκ, Οργάνωση Κοινωνία των πολιτών που δουλεύουν ε, και θα τη φέρουμε εδώ αυτήν την οργάνωση για να μας βοηθήσει ε, να χυθεί άπλετο φω στην υπόθεση αυτή της Ρουμανίας. Ο κύριος Κοέγιο ε, και άλλοι συνάδελφοι τόνισαν ότι δεν θα κάνουμε μία έρευνα εμείς. Πολύ σωστό αυτό, σωστό να το πούμε, για να μην υπάρχει καμία αμφισημία. Ε, ε, δεν είμαστε εμείς Είμαστε εμεί επικεφαλή μια ε, επιτροπή, όπω και εσεί κύριε Κοέγιο. Θα συντάξουμε απλώ μια έκθεση που ελπίζω, μια έκθεση δίας πρωτοβουλία που θα εντοπίζει, ελπίζω, ε, τα εμπόδια ε, στην αλήθεια και στη δικαιοσύνη. Οι Ευρωπαίοι πολίτε χρειάζονται αυτή τη δικαιοσύνη και την αξιοπιστία. Τη χρειάζεται την αξιοπιστία αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. πρέπει και για να είναι αποτελεσματικός ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας. Και υπόθηκε από αυτό το βήμα ότι στις ΗΠΑ αλλά και αλλού ε, περιμένει πολλά ο κόσμος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, περιμένει ε, να παίξει το ρόλο της αιχμής του δόρατος για τη δικαιοσύνη και την αλήθεια. Και αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ όλους για την συνεισφορά σας, για την προσοχή σας. Νομίζω ότι προϊονίζεται μια πολύ καλή δουλειά, μια δουλειά που θα είναι στο ύψος των προσδοκιών που εκφράστηκαν σήμερα το πρωί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρία Φλότχα για τους προβληματισμούς, τις σκέψεις σας. Ε, ολοκληρώνουμε έτσι την πρωινή συνεδρίαση. Και τώρα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές των τριών πάνελ ε, που μίλησαν σε αυτή την ακρόαση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. και μην ξεχνάτε ότι θα είσαστε έμπνευση ε, για, την έκθεση δικής μας πρωτοβουλίας που θα συντάξει η, έκθε, η, η συντάκτριά μας η κυρία Φλότ και ε, της έκθεσης της κυρίας Λάντφορντ ε, αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Άφετη, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα υπάρξει ένα follow-up αυτής ε, της ακρόασης, μια συνέχεια αυτής της ακρόασης, στις 12 Απριλίου. Στην υποεπιτροπή Ντρουά. Και τώρα, περνάμε στην ψηφοφορία. Παρακαλώ, προσοχή. Προσοχή. Θα ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Παρακαλώ λοιπόν ε, ε, σιωπή λίγο γιατί θα ψηφίσουμε και πρέπει να είστε λίγο προσεκτικοί. Παρακαλώ λοιπόν ε, να είστε προσεκτικοί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τις, ψηφολο... με τις ψηφοφορίες στην ώρα μας χωρίς καθυστέρηση. Ε, καταρχήν έχετε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες. Όσοι δεν τις έχουν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 Παρακαλώ λοιπόν τους ευρωβουλευτές, ε, ε, αυτοί έχουν δικαίωμα να κάθονται καταρχήν. Καταρχήν. Οι ευρωβουλευτές έχουν δικαίωμα να έχουν κάποιο κάθισμα για να μπορέσουν να διεκπαιρεώσουν την ψηφοφορία. Δεύτερον, Όσοι δεν συμμετέχουν στην ψηφοφορία παρακαλώ να βγουν από την αίθουσα ή να είναι ε, σιωπηλοί για να μπορέσουμε να συγκεντρωθούμε στην ε, ψηφοφορία και να είμαστε σίγουροι ότι όσοι έχουν δικαίωμα ε, ψήφου πρέπει να έχουν θέση και την ηλεκτρονική τους κάρτα κατά προτέμηση μαζί τους διότι θα γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος των ψηφοφοριών. Εάν τώρα λοιπόν είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν οι προποθέσεις για να συνεχίσουμε, όλοι είναι καθισμένοι, όλοι έχουν τις ε, κάρτες τους, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Είμαστε στο σημείο 9 σύναψη της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τη χρήση και την διαβίβαση των φακέλων επιβατών φάκελοι PNR στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ. Ο εισηγητής ήταν η κυρία Σόφη Ιντβελτ και τώρα θέλουμε να ψηφίσουμε ε, την, ε, το σχέδιο γνωμοδοτήσεως ε, σχετικά με το σχέδιο συμφωνίας για τα PNR μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πρέπει να διευκρινίσω τη διαδικασία. Η ψηφοφορία βάσει του σχεδίου της εισηγητρίας ε, σας υπενθυμίσω τι έγινε στο TFTP ή στη συμφωνία για τα PNR με την Αυστραλία σημαίνει ότι ισχύει το εξής. Ένα, εάν υπερψηφίζεται, ε, αν ψηφίζετε υπέρ σημαίνει ότι καταψηφίζεται τη συνένεση ή τη συμφωνία. Ε, αυτοί που θέλουν να καταψηφίσουν την ε, συμφωνία πρέπει να υπερψηφίσουν το σχέδιο γνωμοδοτήσεως ε, της εισηγητρίας. Αλλά όσοι καταψηφίσουν τη γνωμοδότηση θα υπερψηφίσουν την συμφωνία. Οπότε ε, να το θυμάστε για να μην ε, ε, υπάρξει παρανόηση μπορείτε να κάνετε δήλωση αν θέλετε αν δεν υπάρχουν δηλώσεις παρακαλώ να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία η οποία ξεκινά τώρα ηλεκτρονικά Καταφαινόμενο όμως όχι Υπάρχει ένα πρόβλημα, λέει ο πρόεδρος, με ε, το δικό μου μηχάνημα. Οι φιλελεύθεροι έχουν έναν πλεονάζοντα ευρωβουλευτή ο οποίος ψηφίζει. Λοιπόν, έχουμε δύο σοσιαλιστές πλεονάζοντες και ακόμη έναν. Κάποιος ευρωβουλευτής των σοσιαλιστών πρέπει να βγάλει την ε, κάρτα του. Παραμένει, παραμένει ένας σοσιαλιστής ε, ο οποίος είναι πέραν των επιτρεπομένων. Ο Κλοντ ποιος είναι ο πλεονάζων. Ένα λεπτό ε, θα το ελέγξω. Λοιπόν, μειώθηκε. Όχι, ακόμη. Υπάρχει ακόμη ένας όμως. Να επαναλάβουμε την άσκηση για να δούμε αν τώρα είμαστε όλοι εντάξει. Επαναλαμβάνουμε τη δοκιμαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ε, είχαμε έναν ε, σοσιαλιστή επιπλέον και ξεκινά η ψηφοφορία. Πού βρισκόμαστε? Είμαστε εντάξει. Ωραία. Οπότε λίγη ψηφοφορία. 31 κατά, 22 υπέρ. Ο Οπότε το σχέδιο γνωμοδοτήσεως δεν υιοθετήθηκε αλλά βλέπω ότι ο κύριος Ταβάρες είναι εδώ, δεν έχει την κάρτα του, ψήφισες, ναι. Άρα έχουμε ένα ναι επιπλέον, 23 υπέρ και 31 κατά. Αυτή είναι η τελική καταμέτρηση. Τώρα προχωράμε στην επόμενη ψηφοφορία η οποία είναι πιο περίπλοκη. Now, please. Τώρα. Υπάρχουν διάφορες ψηφοφορίες που μας περιμένουν κάπως πιο περίπλοκες. Συνεπώς, παρακολουθήστε με παρακαλώ. Ψηφίζουμε την ε, πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό που καθορίζει κώδικα για την μετακίνηση των ε, ατόμων ε, Σέγγεν δηλαδή και την ε, σύμβαση εφαρμογή της Συμφωνίας Σέγγεν. Η συγκητής μας είναι ο κύριος Γιώργος Παπα-Νικολάου, ο οποίος δεν χρειάζεται να πάρει το λόγο, αν δεν θέλει. Ψηφίζουμε. Τροπολογία αριθμός 1. Υπέρ παρακαλώ.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 Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική αριθμό 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οπότε καταπίπτουν διάφορες τροπολογίες και φτάνουμε στην 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά γιατί δεν ήταν σαφέ το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 48. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορίες. 20 κα... 29 υπέρ, 24 ε, κατά, εγκρίνεται. 13 τώρα, που είναι συμβατή με την προηγούμενη. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 19 έχει αποσυρθεί, 52 την ψηφίζουμε. 52 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 53 υπέρ. Για να ελέγξουμε. Για την, για την 22 ελέγχουμε. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρες ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε με 27 υπέρ, 24 κατά. Εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. Α, συγγνώμη, απορρίπτεται ήθελα να πω. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλα, ψηφίζουμε. Για την 25 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. 25. τη πληροφορία. Υπάρχει κάτι που δεν λειτουργεί. Α, εγκρίνεται, εγκρίνεται, ναι. Συγγνώμη, εγκρίνεται, λέει ο πρόεδρο. Σαφώ με 55 υπέρ. 56 τώρα υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. απόχέ Για να ελέγξουμε. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 26 παρακαλώ. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα στις ψηφοφορίες. 27 υπέρ, 28 κατά. Απορρίπτεται. 57 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 58 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Εγκρίνεται, εγκρίνεται ήθελα να πω διορθώνει ο πρόεδρος. Εγκρίνεται, ναι. Όχι, δεν χρειάζεται να ελέγξουμε, ναι. Λάθος, το είπα. Εγκρίνεται. 30 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε τώρα. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 30. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της προφοριες 27 27-29 απορρίπτεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω. Αλλά να ελέγξουμε γιατί 33. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. 24 υπέρ 30 κατά απορρίπτεται. 34 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 63 έχει αποσυρθεί και 24 και 25 και 26. Πάμε στην 35. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω. 67 έχει αποσυρθεί. 68 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 60 έχει αποσυρθεί. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Κάποιες καταπίπτουν και πάμε έτσι στη συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάλι εδώ κάποιες καταπίπτουν και πάμε στην 37 υπέρ παρακαλώ κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας της ψηφοφορίας, 36 υπέρ, 20 κατά. Εγκρίνεται. Έτσι πάμε στην τροπολογία αριθμός 38. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 39 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 40. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται νομίζω. 74 είναι συμβατή με την 40, άρα πρέπει να την ψηφίσουμε. 74. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 76. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της προφορίας. 29 υπέρ, 27 κατά. Εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε. 78 ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας 29 υπέρ 27 κατά εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ κατά αποχές πάλι θα ελέγξουμε για την 80 ηλεκτρονικά ψηφίστε πέρα στις Η 28 28-28 είναι το αποτέλεσμα άρα απορρίπτεται ναι βλέπω να το χέρι ναι το βλέπω ε, εντάξει Ε, εντάξει, ναι. Το καταλάβαμε. Κερδίσατε. 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 81 κατά, αποχές απορρίπτεται. Τώρα περνάμε σε τριλογικές σκέψεις και προτάσεις. Πρώτα απ' όλα τροπολογία 43 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 44 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα τροπολογία 7 είναι γλωσσική τροπολογία και ε, προχωράμε στο κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί ηλεκτρονικός έλεγχος. Ξεκινά η ψηφοφορία ηλεκτρονικά, λίγη. 51 υπέρ, 3 κατά και 2 αποχές, δηλαδή ενεκρίθη. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπα-Νικολάου. Και προχωράμε στην τρίτη ψηφοφορία η οποία είναι επίσης περίπλοκη. Είναι αρκετά μακριά. Εδώ ψηφίζουμε την πρόταση για μια οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την φορολόγηση των συστημάτων πληροφοριών και κατάργηση της απόφασης η οποία ε, είχε ε, ε, για τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών και κατάργηση της απόφασης σχετικά του Συμβουλίου. Παρακαλώ προσοχή για να μην ξεπεράσουμε το χρόνο μας. Πρέπει δηλαδή ουσιαστικά στις 12.30 να ολοκληρωθεί η ε, ψηφοφορία και πρόκειται για μια περίπλοκη ε, ψηφοφορία. Η κυρία Χολμάγερ που είναι συγγήτρια ε, θέλει τον λόγο. Όχι, δεν χρειάζεται. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, την κυρία Χολμάιερ η οποία μας εξοικονόμησε χρόνο με τις ε, εσωτερικές παρατηρήσεις. Συμβιβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το 75 απεσύρθη συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το 17 απεσύρθη, τα υπόλοιπα καταπίπτουν, το συμβιβαστική 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ορισμένες έχουν καταπέσει, η συμβιβαστική, η τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προχωρούμε στη συμβιβαστική 17 υπέρ. Κατά αποχές ε, συμβιβαστική μάλλον όχι, τροπολογία 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μέχρι την 93 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 έχει, ε, έχει καταπέσει όχι πρέπει να ψηφίσουμε την 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ όχι έχει καταπέσει 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ήτρε 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 ήτρε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ήτρε 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 98 καταπίπτει ή 26 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται καταπίπτει η 99 και η 100 το ίδιο ισχύει και για την 101 αλλά 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Καταπίπτουν οι 103, 104, συμβαστική 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και μία, μία μακριά λίστα τροπολογιών αποσύρονται, καταπίπτουν κατά αυτόν τον τρόπο μέχρι την 118 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές ας ελέγξουμε σχετικά με το δεύτερο τμήμα της 118. Ε, ψηφίζουμε υπέρ. Ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Έληξε. 27 υπέρ, 28 κακά, κατά. 28 με 28 και πάλι ε, ε, απερίφθη. 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 121 υπέρ κατά απορρίπτεται 122 Απορρίπ, ε, αποσύρεται κύριε ναι Ήτρε 23 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται συμβασμός 21 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Μία ολόκληρη λίστα από τροπολογίες καταπίπτουν και πάμε στην 32 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. Άφετ 21 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 127 με προφορική τροπολογία δεν υπήρχε στον κατάλογο η προφορική τροπολογία. Προφορική τροπολογία της κυρίας Βεργιά, παράγραφος 2. Υπάρχει στον κατάλογό σας, δεν υπήρχε στο δικό μου, συγγνώμη, γι' αυτό έκανα το λάθος. 127 υπέρ, κατά, εποχές, Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 127 με την προφορική τροπολογία. Πέρας ψηφοφορίας. 31 υπέρ, 22 κατά. Υιοθετείτε. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33 υπέρ. Against abstentions adopt. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Ήτρε 27. Διορθώνει μιλτής Ήτρε 28. Υπέρ. Κατά. ποχές, υιοθετείτε. Τώρα, αιτιολογικές σκέψεις και αναφορές. Η συμβασμός 1. Υπέρ. Κατά. ποχές, υιοθετείτε. Ήτρε 2. Υπέρ. Κατά. ποχές, υιοθετείτε. Συμβασμός 2. Υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείτε. Φεύγουν διάφορες και πάμε στην ήτρα 4 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείτε. Ήτρα 5. Λάθος κάνω. Λάθος. 38 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείτε. Συγγνώμη κύριε Ενσιού που ήταν και δική σας τροπολογία. Ήτρε 5. Υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείτε, ή 6 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται άφετ 5 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται άφετ 6 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται συμβιβάσμος 3 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται ήτρε 8 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 44 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 3 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 4 η προηγούμενη του Axel έχει ήδη καλυφθεί. Πάμε στην τροπολογία 4 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 5 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 6 υπέρ, κατά, εποχές, υιοθετείτε. Κάποιες καταπίπτουν, κάποιες έχουν αποσυρθεί, καταπίπτουν και όμως 48, υπέρ, κατά, εποχές, υιοθετείτε. Τι πήδηξα. Ο συμβασμός 5 έχει ψηφιστεί. Και η 48 έχει ψηφιστεί ήδη. Ήτρε 12. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείτε. Άφετ 10. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείτε. Συμβασμός 6. Συμβασμός 6 υπέρ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείτε. Ήτρε 13 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 8 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. Ήτρε 14 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. Άφετ 12 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. Συμβασμός 7. Το ψηφίσαμε. Όχι, πρέπει να το ψηφίσουμε. Υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Κάποιες καταπίπτουν. Πάμε στο συμβασμό 8. Υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείτε. Κάποιες από τις επόμενες καταπίπτουν. Κάποιες έχουν αποσυρθεί. Συμβασμό 9 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. Κύριε Φλασίκοβα επίδειξα κάποιο αιτιολογική σκέψη. Δεν φτάσαμε ακόμα εκεί που λέτε. Συμβασμό 9 υπέρ. Τροπολογία 11. Έχει αποσυρθεί. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβασμός 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Αποξίωτη επόμενη. Καταπίπτουν οι άλλες. 11. Συμβασμός 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 12. Συμβασμός 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. 68. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Ο συμβασμό 13 καλύπτει μερικές από τι επόμενε και πάμε στην 71. Όχι, την 70. Με προφορική τροπολογία. 70 με την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. Ελέγχουμε Ψηφίζουμε. 71. Πέρας. 24 υπέρ, 29 κατά. Απορρίπτεται. Άφετ. 15 υπέρ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείται. Άφετ 16 υπέρ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείτε. Ψηφίζουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζεται. Πέρας ψηφοφορίας. 50 ε, υπέρ, 3 αποχές, μία ψήφος κατά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς που μας δίθεσαν λίγο παραπάνω χρόνο. Έκαναν υπερορία. Γεια σας.